Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να συνεχίσουμε με την συνεδρίαση μας. Είναι μεγάλη μου τιμή, όπως πάντα, που έχω την ευκαιρία να αποδεχτώ εδώ τον συνηθισμένο μας επισκέπτη, τον κύριο Ανδρής Πίμπαλξ, που είναι Επίτροπος για την Ανάπτυξη. Στόχος της σημερινής μας συνάντησης μαζί του είναι να έχουμε το διαστρωμένο ετήσιο διάλογο επί του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως υπενθύμησα και χτες, στόχος του διαστρωμένου διαλόγου φέτος ήταν πιο διευρυμένος προκειμένου να υπάρξει και αξιολόγηση των πρωτοβουλειών που πήρε η τρέχουσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς ο κύριος Πίβαλξ μπορεί λίγο να μείνει μαζί μας σήμερα, μισή ώρα μόνο και γι' αυτό του δίνω ευθύ αμέσω το λόγο για να μας κάνει μια σύντομη εισαγωγή για πέντε λεπτά περίπου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι εδώ για τον ε, ε, ε παραδοσιακό ε, ε, δομημένο μας διάλογο για να ε, συζητήσουμε τις εξελίξεις και τις προτεραιότητες μας για το 2020. Να σας διασφαλίσω καταρχήν ότι δεν θα χαλαρώσουν καθόλου οι προσπάθειές μας ε, να βελτιώσουμε ε, την αποτελεσματικότητα της αναπτυσιακής ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό στόχος μας θα είναι η εφαρμογή της, του θεματολογίου για αλλαγή που εξακολουθεί να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει και Έχουμε δύο πυλώνες, ε, την ε, αναπτυξιακή ε, ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση, την αναπτυξιακή συνεργασία και, τη διακυβέρνηση. Έχουμε λοιπόν κοινά προγράμματα με περισσότερες χώρες εταίρους. Τώρα καλύπτουμε σχεδόν 40. Οι νέες κατευθυντήρες γραμμές μας οδηγούν σε μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Έχουμε ε, τις ε, τριπλάσιες συμβάσει ε, και έχουμε ενισχυμένα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη διαφάνεια και την εποπτεία. Οι καινοτόμοι, οι οικονομικοί μηχανισμοί μας διαμορφώνονται και θέλουμε να φτιάξουμε ένα ισχυρό πλαίσιο για τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, έχουμε παγκόσμια κάλυψη όσον αφορά τους μηχανισμούς συνδυασμού επιχορηγήσεων και δανείων. Και για το προγραμματισμό μας ε, για το διάστημα 2014-2020 ε, ε, βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που με φέρνει στο θέμα του στρατηγικού διαλόγου και των κατεξουδότηση πράξεων. Οι κατεξουδότηση πράξεις θα δώσουν στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την δυνατότητα να καθορίζουν συγκεκριμένες προτεραιότητες ανά περιοχή. Ο στρατηγικός διάλογος Όσον αφορά τον ε, δεδομένο διάλογο, ε, θα ε, υποβάλω στο Κοινοβούλιο πρόταση κατανομής και δαπάνης των χρημάτων. Θα έχουμε τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και έτσι θα επηρεάσετε τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Πιστεύω ότι η προσέγγιση αυτή μπορεί να μας βοηθήσει να αποφύγουμε Καθυστερήσει ε, στην εφαρμογή της αναπτυξιακή βοήθεια, ε, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε ε, στις ανάγκες. Η εφαρμογή του θεματολογίου για αλλαγή θα συνεχίσει να καθορίζει τις προτεραιότητές μας τα επόμενα χρόνια. Το 2014 μεταξύ άλλων θα συμβάλλουμε σε πιο ισχυρό ιδιωτικό τομέα ώστε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Όσον αφορά την χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Θα συνεχίσουμε τη διετή μας προσέγγιση, να επιταχύνουμε τις ε, υπάρχουσες υποχρεώσεις ε, και να συμμετέχουμε επικοδομητικά στον ε, διεθνή διάλογο. Επίσης, στην ανακοίνωση της Κομισιόν μιλάμε για αξιοπρεπή ζωή για όλους, όπου παρουσιάζουμε ένα εφικτό όραμα ε, και θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω την ε, θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εξετάζοντας τα αποτελέσματα των στόχων της χιλιετίας και με προετοιμασία το 2050 χάρη σε αίτημα του Κοινοβουλίου και της ΕΟΚΕ, ο πρόεδρος Παρόσο συμφώνησε ε, να προτείνει το 2015 να είναι το, διεθνές, ε, το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να δείξουμε την δέσμευσή μας για την καταπολέμηση της φτώχειας σε όλο τον κόσμο και να βοηθήσουμε οι πολίτες να έχουν καλύτερη κατανόηση των αρχών και στόχων και αποτελεσμάτων της αναπτυξιακής συνεργασίας μας. Επίσης, για το 2015, ε, επίσης το 2015 θα είναι μια προθεσμία εξέτασης των αποτελεσμάτων των στόχων της χιλιετίας. Έτσι λοιπόν το 2015 ε, πιστεύουμε ότι θα είναι ε, μια μοναδική και ζωτική σημασία χρονιά για την αναψυχική συνεργασία και αυτό είναι ο λόγος που δεν μπορώ να μείνω όσο θα ήθελα στην Επιτροπή σας ε, διότι η τελική έκθεση του πάνελ υψηλού επίπεδου θα συζητηθεί αύριο και θα πρέπει να υποβληθεί στον Γενικό Γραμματέα την Πέμπτη. Και αυτός είναι ο λόγος που έχω τόσο περιορισμένο χρόνο. Λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Αλλά ε, θα ε, αποζημιώσω το Κοινοβούλιο γι' αυτό όποτε θεωρήσει ότι είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Κόρτες Λάστρα. Δύο λεπτά, καθότι έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο. Δύο λεπτά ο καθένας σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος γιατί και εγώ πρέπει να φύγω. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο για την εισαγωγή του και για τα όσα μας εξήγησε. Του χρόνου θα είναι η χρονιά όπου, 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα κληθούν να ψηφίσουν. Και θα αναρωτηθούν βέβαια τι γίνεται με την ε, συνεργασία μας και γιατί τα μέσα είναι πιο συντηρητικά από ό,τι τα κατά το παρελθόν. Η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ένα πλόκο, δεν φαίνεται να ευνοεί την βοήθεια προς τους ε, πιο φτωχούς. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Δεν είναι δυνατόν ο Επίτροπός μας να αφιερώνει την ομιλία του στην οικονομική ανάπτυξη ενώ πρέπει να επικεντρωθεί και να προσέξει αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη. Δεν είναι δυνατόν να λέγονται συγχρόνως ότι το κλειδί είναι η εργασία και ο ιδιωτικό τομέα. Η ανάπτυξη δεν επιταχύνεται βόβο μόνο με βοήθεια. Χρειάζεται βιώσιμη ανάπτυξη και σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Όμως με τι τίμημα. Γι' αυτό κύριε Πίβατς βλέπω στο πρόγραμμα για το 2014 ένα μεγάλο κενό. Μία πρόταση στρατηγικής που αναφέρει τον ιδιωτικό τομέα και λέει ότι δρά για την κατάργηση της ένδιας και καθορίζει ένα πλαίσιο με δράσεις από τη, που μπορεί να υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διάφορες χώρες με τον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας όμως υιοθετεί έναν, ένα μοντέλο όπως γίνεται και στην Κίνα. Χρειάζεται μια στρατηγική με όραμα για το μέλλον και να έχει τη θέση του στην ανάπτυξη, αλλά η ανάπτυξη να καθορίζεται συγκεκριμένα και να συνάδει με τις δικές μας αρχές και αξίες. Μια στρατηγική που να αναγνωρίζει την ανάγκη ενός ισχυρού ιδιωτικού τομέα της υπονάπτυξη χώρας, αλλά συγχρόνως να δίνει ένα όραμα για το ρόλο των ε, επιχειρήσεων που να είναι όπως πιστεύουμε εμείς. Και ολοκληρώνω. Κύριε Μίτσελ, η σειρά σας. Έχετε το λόγο κύριε Μίτσελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Thank you, for... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη για την μικρή μου καθυστέρηση. Ε, ήμουν σε συναευρίαση με τον πρόεδρο της Επιτροπής και τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Σε σχέση με το 2014 και την σχετική, τα σχετικά προγράμματα, συγγνώμη, του 2013, ε, και τα ζητήματα δηλαδή τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε φέτος και του χρόνου, πιστεύω ότι θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα ε, σε ένα συγκεκριμένο, στη δημιουργία ενός συγκεκριμένου ταμείου ε, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κακής διατροφής, της ελληπούς διατροφής. Δεν είναι δυνατόν να ε, δεχτούμε μια κατάσταση ε, όπου εκατομμύρια είναι οι γυναίκες οι οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους και χιλιάδες, είναι 200.000 κάθε χρόνο, οι οποίες δεν μπορούν να τραφούν σωστά. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Χαίρομαι γιατί η Επιτροπή παίρνει περισσότερα ενεργά μέτρα όσον αφορά ε, την αντιμετώπιση κακών ε, καταστροφών και ε, ειδικών καταστάσεων. Νομίζω ότι εάν βάλουμε 3 ευρώ σε αυτό το Ταμείο Προστασίας και Πρόληψης των Καταστροφών ε, θα κερδίζουμε για κάθε 3 ευρώ 12 ευρώ. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν και άλλα δύο ε, σημεία όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ενισχυμένη συμπληρωματικότητα ε, ε, δημιουργώντας ένα κοινό, ε, μια κοινή προσπάθεια. έξι δις κάθε χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν, να εξοικονομηθούν μάλλον. Επίσης πέρα από, την, ε, από τις διαφορές των φίλων, γιατί ε, υπάρχει ε, πάντα η εντύπωση ότι οι άντρες είναι αυτοί οι οποίοι οδηγούν την οικονομία και έχουν μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια αλλά πρέπει να προωθήσουμε όλες τις επιχειρήσεις. Ο κύριος Γιώνας για δύο λεπτά και δεν θα τα ξεπεράσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να σας πω τα συγκεκριμένα μου σημεία. Πρώτον, συνοχή και πολιτική. Μας λένε ότι η Κομισιόν μέχρι το Σεπτέμβριο οπωσδήποτε θα ε, ε, παρουσιάσει έκθεση και όχι ανακοίνωση όσον αφορά την συνοχή μεταξύ των πολιτικών. Νομίζω, όπως κατάλαβα, ότι η έκθεση ε, είναι πιο ε, χαμηλής θεσμικής ε, πυκνότητας και σημασίας από την ανακοίνωση. Όμως θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο γιατί η συνοχή των πολιτικών για τα θέματα που μας απασχολούν είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερο θέμα, η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κύριος πρωταγωνιστής ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας. Νομίζω ότι και η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχουν μεγάλη ευθύνη. Σήμερα ε, συζητούσαμε το θέμα της ένταξης των, της βιομάζης ε, εις τα καύσιμα ε, και είπαμε ότι βεβαίως δεν θέλουμε να υπάρχει λαιλασία των φυσικών πόρων των αναπτυσσόμενων χωρών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να ισχύσει μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της δεν είναι οι μόνες οι οποίες δρούν επιτόπου και οι εταίροι μας ε, και οι άλλοι οι οποίοι δρούν επί τόπου θα πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Ε, και βεβαίως ε, μέχρι το τέλος της νομοθεσίας, η νομοθετική μας εργασία επ' αυτού έχει ολοκληρωθεί. Γι' αυτό θα ήθελα να μας πείτε κάτι. Τρίτον, Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Βουκ Τζέρεμιτς, ο οποίος είναι πρόεδρος της Συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών. Έμαθα λοιπόν ότι υπάρχουν τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων τρεις ε, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία, δηλαδή οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν εμπλακεί στη διαδικασία προετοιμασίας ε, για την, ως, ως διαμεσολαβητές ε, για την οργάνωση του συνεδρίου για την ανάπτυξη. Εκτός από τις τρεις χώρες υπάρχει και η Νορβηγία, η οποία ξέρουμε ότι δεν είναι πολύ ανοιχτή για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ο κύριος Πίπα για, για ε, δύο λεπτά επίσης και μετά θα έχουμε ένα δεύτερο ε, γύρο. Well, uh, uh, to Mr. Στον κύριο Κόρτες Λάστρα να πω ότι σίγουρα η φτώχεια είναι βασικό επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας, ε, αλλά αν, ακολουθήσετε, αν παρακολουθείτε τη συζήτηση στην Αφρικανική Ένωση εδώ και 50 χρόνια, θα διαπιστώσετε ότι ε, οι χώρες ε, θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να αντιμετωπίσουν μόνο του τη φτώχεια. Για να είναι αλήθεια αυτό όμως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, κάποια συγκεκριμένα προβλήματα και έχουμε ασχοληθεί με την ασφάλεια παροχής τροφίμων και άλλα. Πρόκειται λοιπόν για επενδύσεις ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στις χώρες να ξεφύγουν από τη φτώχεια και για τον ιδιωτικό τομέα. Νομίζω ότι είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει εδώ δυναμικό, διότι ε, δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Αν δώσουμε τη δυνατότητα ε, στον ιδιωτικό τομέα να αναπτυχθεί, τότε αυξάνουμε τη δυνατότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι... Λοιπόν, η βασική μας στόχη, αλλά πρόκειται για εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια. Όσον αφορά την ερώτηση του Γκέι Μίτσελ, ε, το Trust Fund για τον υποσυτισμό, ε, ειδικά στην Αφρική, ε, θέλουμε να ενισχύσουμε την αντίσταση στις φυσικές καταστροφές. Γι' αυτό η διατροφή θα είναι σημαντικό ενδιαφέρον μας και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ε, ακολουθήσουμε αυτήν την ε, γραμμή. Θα εξετάσουμε το θέμα των τράσφαντα, αλλά πιστεύουμε ότι η διατροφή και ότι τα οχήματα, τα ηλιακά οχήματα, επίσης θα πρέπει να συνεχίσουν να μας αποσχολούν. Επίσης, ε, Όσον αφορά το πλαίσιο αποτελεσμάτων θα ετοιμάσουμε έγγραφο και όσον αφορά τον κύριο προγραμματισμό προοδεύουμε σε 40 χώρες έχουμε σημαντική πρόοδο ε, για να πετύχουμε τα 6 δισεκατομμύρια, αλλά πιστεύουμε ότι μπορούμε να εξοικονομήσουμε ακόμα περισσότερα. Όσον αφορά την ερώτηση του Charles για το PCD, ε, θα εξετάσω αυτό που λέτε. Για μένα η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, όσο και η επικοινωνία. Γι' αυτό σημαντικό για μένα είναι να έχουμε εδώ την σωστή προσέγγιση. Τον Οκτώβριο ε, προβλέπουμε την έγκρισή του. Ε, λυπάμαι λίγο που καθυστερούμε τόσο, έτσι με ενημέρωσε το προσωπικό μου, αλλά ε, πιστεύουμε ότι αυτό είναι σημαντικό, να υπάρχει δηλαδή πολιτική συνοχή για την ανάπτυξη. Για την ανάπτυξη. Επίσης, ε, επικεντρωνόμαστε σε δύο πράγματα, το ε, πλαίσιο μετά το 2015 και το άλλο που θα έχουμε την πρώτη υπουργική συνάντηση μάλλον φέτος και ε, η Νιγηρία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ινδονησία ε, θα ηγηθούν στι εργασίε αυτέ. Ελπίζω ότι θα λειτουργήσει καλά και όσον αφορά τον συντονισμό των προσπαθειών μα. Ε, προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με όλου που έχουν ίδιε απόψει με εμά και να βρίσκουμε χορηγού. Ευχαριστώ πολύ. Η σειρά μου για δύο λεπτά. Και εγώ. Χτες η Επιτροπή Ανάπτυξης είχε μία ακρόαση για το θέμα του blending, δηλαδή της συνδυασμένη χρηματοδότησης. Θα θέλαμε να έχουμε και ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό, προκειμένου να μπορέσουμε τελικά να καταλήξουμε στην άποψή μας, να διαμορφώσουμε άποψη. Στην αρχική ακρόαση μας είχατε υποσχεθεί να εντοπίσετε τα κράτη-μέλη τα οποία δεν τιμούν τις υποχρεώσεις τους να πληρώνουν 0,7% του έπτους. Τελικά, τι κάνατε προκειμένου οι χώρες αυτές να τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Είπατε επίσης ότι δεν είναι δυνατόν να μπορούμε να βοηθήσουμε τις χώρες άμα από την άλλη μεριά τους κλέβουμε τους φυσικούς τους ε, πόρους. Αυτό όμως συμβαίνει δυστυχώς και δεν έχουμε δει καμία αντίσταση. Είδαμε επίσης ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης ε, θέλουμε να προχωρήσουν ακόμα και αν είναι κατά οι χώρες ΑΚΕ και πιέζουμε. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την αντίφαση, πώς την αναλύετε και τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε ώστε να μην μπορέσετε να έχετε κάνει κάτι μέχρι τώρα. Συγχρόνως διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει συνοχή όσον αφορά την ανάπτυξη. Υποσχεθήκατε ότι θα συντονίζατε την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώνουμε όμως με τη Σιμπάμπουε, τη Μαδαγασκάρη, ότι προχωρούν οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου χωρίς πραγματικά αν υποστηρίζονται τα συμφέροντα των χωρών αυτών. Υπάρχει δηλαδή σύγκρουση συμφερόντων εδώ. Εσείς προσωπικά τι κάνατε λοιπόν για να διασφαλίσετε ότι το άρθρο 208 της συνθήκης τηρείται και υπάρχει συνοχή στην πολιτική μας αυτή. Η κυρία Σαρτζεντίνη είναι η επόμενη. Ευχαριστώ. Στον πρώτο γύρο απαντήσεων άκουσα τον Επίτροπο να λέει ότι ο ιδιωτικός τομέας και τα ανθρώπινα δικαιώματα πάνε μαζί. Και είπατε ότι μια επιχείρηση θα επενδύει σε μια χώρα μόνο εφόσον υπάρχει κράτος δικαίου και υπάρχει και μια επενδυτική νοτροπία ασφαλής. Ωραία, σωστό. Όμως, Αυτό το κράτος δικαίου και αυτή η ηρεμία, η ηρεμία, το καλό επενδυτικό κλίμα, πώς έχει εγκαθιδρυθεί. Εδώ εμεί συζητούμε για το εμπόριο και την αναπτυξιακή πολιτική και πολλές φορές ο κόσμος καταλήγει να πιστεύει ότι τελικά είναι οι επιχειρήσεις αυτές που επιβάλλουν το κράτος δικαίου, το δικό τους δίκαιο ουσιαστικά. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι οι χώρες θα πρέπει να συνεργάζονται. Οι χώρες δηλαδή που παίρνουν αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει εκείνες να δημιουργούν το κράτος δικαίου πρώτα και τους δημοκρατικούς θεσμούς και μετά να γίνονται οι επενδύσεις αυτές από τον ιδιωτικό τομέα. Αν δούμε τη συζήτηση που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα ODAs, είμαστε κάτω από το 0,7% αναπτυξιακή βοήθεια. Και τελικά η συζήτηση γίνεται περισσότερο για το εμπόριο και όχι για τη βοήθεια. Trade, not aid. Οπότε και η Επιτροπή μας, αλλά και εσείς που είσαστε για την αναπτυξιακή συνεργασία, πρέπει να ξαναδούμε τελικά τη θέση μας. Να υπάρχει συνοχή ε, με την ανάπτυξη και σε όλες τις πολιτικές να εξετάζουμε το θέμα της ανάπτυξης. Μας έδωσε ένα παράδειγμα η Πρόεδρος και θα σας δώσω κι εγώ ένα άλλο παράδειγμα. Η δυνατότητα για την πρόταση de για ένα ελάχιστο στην νομοθεσία. Το εξετάζει αυτή την εποχή και ελπίζει πριν τα Χριστούγεννα να μπορέσει να έχει δημοσιεύσει κάτι. Ελπίζω να μπορέσω να το υποστηρίξω, αλλά από πλευρά αναπτυξιακή. πώς θα διασφαλίσουμε ότι έχουμε βιώσιμη εξόριξη. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο για να απαντήσετε και για να ολοκληρώσουμε την ανταλλαγή αυτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το blending, αυτό το μείγμα θα το λάβουμε υπόψη μας, αλλά θα, θα προετοιμάσουμε και επιπλέον επεξηγήσεις προς το Κοινοβούλιο, έτσι ώστε ε, να, ε, ώστε να ε, δούμε ακριβώς τι εννοούμε με το blending. Δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι η βοήθεια η οποία δίνεται μέσω των, του Ταμείου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς επίσης και μέσω των επενδυτικών το μείγμα για της Επενδύσεις. Ε, βεβαίως κατανοώ ότι υπάρχει δυστημία όσον αφορά τα επιτεύγματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ που θεωρώ, κυρία Πρόεδρε, ότι ό,τι υποσχέθηκα το έκανα. Το 0,7% είναι το συμπέρασμα ε, του, τον, ε, είναι η κατάληξη μάλλον ε, του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Αλλά εγώ λέω ότι ακόμα και σε μια εποχή όπου η πολιτική εστίαση δεν αφορούσε αυτό το θέμα, καταφέραμε και διατηρήσαμε αυτό το ποσοστό. 0,7% ακόμα και για χώρες όπως η δική μου που δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο να ε, πιστούν στο Συμβούλιο αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε saying that it is betraying European citizens. We change the language. Ε, σκληρή γλώσσα γιατί λέμε ότι δεν μιλάμε μόνο για κινδύνους, δεν μιλάμε μόνο για αλληλεγγύη, ε, ε, μιλάμε για την διασφάλιση της στοιχειωδών αναγκών που συνεπάγονται την ασφάλεια των πολιτών, την ασφάλεια της εργασίας, την ανάπτυξη κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Βεβαίως ε, μπορεί κανείς ε, να πει ότι ε, η ανάπτυξη που είναι 0,73% μπορεί να είναι χαμηλό, αλλά οπωσδήποτε θα αυξηθεί και πιστεύω ότι και από την πλευρά της Κομισιόν πιέζουμε και προχωράμε προς σωστή κατεύθυνση. Τώρα, ε, όσον αφορά τα εργαλεία για την ανάπτυξη, πολλές προτάσεις ε, ε, έγιναν, αλλά νομίζω ότι η πιο καλή και η πιο διαφανής ήταν η πρόταση του Επιτρόπου Μπαρνιέ, η οποία κατά την άποψή μου αποτελεί και ορόσημο στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα της ε, ε, φόρο διαφυγής ε, ήταν όντως πάρα πολύ σημαντικό και βλέπω ότι έχουν γίνει πολλές πρόοδοι και μάλιστα στην κορφή της ατζέντα και με το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται το θέμα αυτό. Όσον αφορά το land grabbing ε, και εκεί έχουμε εκδώσει κατευθυντήριες ε, γραμμές για την αηφόρο κάλυψη των αναγκών των καλλιεργητών και την κάλυψη των αναγκών ε, διατροφής κυρίως για τους μικρούς γεωργούς, για τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Νομίζω ότι και εδώ έχουμε ένα αρκετά ικανοποιητικό ε, αποτέλεσμα για τα ε, EPA. Κοιτάξτε, κανένας δεν μας ε, λέει ακριβώς και καθαρά πού δεν πάει καλά αυτό το σύστημα. Ε, τουλάχιστον τώρα αναφέρονται και από τους αρμοδίους επιτρόπους κάποια συγκεκριμένα θέματα που δεν πιστεύω ότι μπορούν να εμποδίσουν τις εμπορικές ε, συμφωνίες. Βεβαίως θέλουμε ένα ε, ε, καθαρό περιβάλλον, βεβαίως θέλουμε καθαρές διαδικασίες ε, που θα ανταποκρίνονται και στις ε, αρχές ε, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. και δεύτερον ε, όσον αφορά την περιφερειακή ολοκλήρωση ε, στην ε, Αφρική μονάχα 10% επιτυχία υπάρχει εδώ και νομίζω ότι αυτό εμποδίζει την Αφρική να αναπτυχθεί και περισσότερο. Όταν μιλάμε με τους εταίρους μας, τους προσπαθούμε να τους κάνουμε να μας μιλήσουν καθαρά. Δεν τους κάνουμε κήρυγμα, θέλουμε να ε, μας πούν ακριβώς τι δεν τους αρέσει. Και ο Επίτροπος δεγούχτο το ίδιο έκανε, προσπάθησε να πιέσει έτσι ώστε να έχει συγκεκριμένε απαντήσεις και αν θέλετε να κάνετε κάποια πρόταση να την ε, ακούσουμε και να την υλοποιήσουμε. Γιατί χωρίς προτάσεις δεν μπορούμε και εμείς να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε. Πάντως θεωρώ ότι η κατάσταση γενικά έχει βελτιωθεί. Και η τελευταία έκθεση σαφώς δείχνει ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα επιτυχίας και πρόοδου μάλλον από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όσον αφορά ε, και θέματα γεωργίας και θέματα μετανάστευσης ε, έχουμε, έχουμε σημαντικές ε, πρόοδους αλλά βεβαίως εξαρτάται και πώς βλέπει κανείς το ποτήρι μπορεί να το βλέπει κανείς μισοάδιο ή άλλος μισογεμάτο εμείς προτιμούμε να λέμε ότι το ποτήρι είναι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο Τέλος δυνατότητα αντίδρασης σε καταστροφές και σε σχέση με αυτό που συνέβη στο Μπαγκλαντές. Σαφέστατα, ρητά είπε η Κομισιόν ότι δεν το δεχόμαστε αυτό και ε, έχουμε ενισχύσει την ε, συνεργασία μας, όχι μόνο με τον Παγκλαντές αλλά και με άλλες χώρες, έτσι ώστε ε, να πλησιάσουν περισσότερο στα δικά μας πρότυπα και να έχουν κοινωνική ευθύνη. Ε, και εγώ και εδώ, και εδώ θέλω διαφάνεια πιστεύω και εγώ ότι η διαφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Ήταν φιλόδοξο το πρόγραμμα του Επιτρόπου και η πρόταση του Επιτρόπου ε, Μπαρνιέ και είμαι σίγουρος όμως ότι το καινούργιο πρόγραμμα θα είναι ακριβώς το ίδιο φιλόδοξο και θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο που ήταν μαζί μας σήμερα και που απάντησε στις ερωτήσεις μας. Την επόμενη φορά είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας μαζί του. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Pour les votes, on n'est pas nombreux. Oui.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 Συνεχίζουμε με τη συνεδρίασή μας και περνάμε στη ψηφοφορία. Σας παρακαλώ ετοιμάστε τις κάρτες ψηφοφορίας γιατί θα κάνουμε μια δοκιμή τώρα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ ενδεικτικά. Ψηφίσατε. Δοκιμάζουμε, κάνουμε δοκιμή για την ψηφοφορία, να δούμε αν όλα λειτουργούν κανονικά. Άλλοι 7 πρέπει να ψηφίσουν. Βάλτε τις κάρτες σας δοκιμαστικά. Κοντεύουμε. Άλλοι δύο Ένας μένει που δεν έχει ψηφίσει. Α, πέρα στις φοφορίες. Ωραία, ψηφίσατε όλοι. Καλώς. Ψηφίζουμε πρώτα τους αλληλευτικούς περιορισμούς και χωρικά ύδατα στη Μεσόγειο για τον εύξενο πόντο. Τρόπο επίλυσης συγκρούσεων. Συμβιβασμός Α. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά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 αποχές εγκρίνεται. Η ηλεκτρονικά τώρα θα ψηφίσουμε. Ψηφίστε παρακαλώ με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Ωραία, εγκρίθηκε ομόφωνα. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Πού είμαι εγώ λέει Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, πρωτόκολλο της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τη δίκαια και ισότιμη συμμετοχή στο φέλη. Δεν υπάρχουν τροπολογίες εδώ, ψηφίζουμε την ε, γνωμοδότηση ως έχει. Υπέρ παρακαλώ κατά εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά, τώρα ψηφίστε. Πέρα της φοφορίας. Ομόφωνα. Συγχαρητήρια στο, στη συντάκτρια την κυρία Γκρέσ που δεν είναι όμως εδώ. Τώρα ψηφίζουμε την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και δίκαιη και ισότιμη συμμετοχή στα ωφέλη που προκύπτουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση. Εδώ έχουμε πολλές τροπολογίες. Τροπολογία 27 υπέρ, κατά αποχές. Μαζί να τις ψηφίσουμε, αν μπλοκ, όχι, εγκρίνεται, καλώς. Δεν μπορούμε ούτε μερικές, όχι, καλά, 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε. Τροπολογία 29. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Τροπολογία 34. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι. Καλά, θα ελέγξουμε. 35. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας της φοφορίες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μέχρι και τη 41 μαζί, 39, 40, 41. Ψηφίζουμε μαζί τις τρεις αυτές τροπολογίες. Σύμφωνοι. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μαζί μέχρι και την 49. Τροπολογία 44 με 46 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κύριε Γκέρενς, θέλετε το λόγο. Όταν έχουμε τροπολογίες που ο συντάκτης προτείνει, νομίζω ότι μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Εδώ είναι καμιά δεκαριά τέτοιες, η μία μετά την άλλη. Δεν μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. Ας προσπαθήσουμε, έτσι κερδίζουμε χρόνο, με τι άλλο. Είναι της ίδιας της συντάκτριας της νομοδότησης. «53 με 56 λοιπόν, υπέρ» κατά, αποχές εγκρίνονται. 57 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 86 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 86 θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Άλλος ένας πρέπει να ψηφίσει. Πέρα της ψηφοφορίες. Απορρίπτεται.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 Τροπολογία 88 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 73 με 79, 73 με 79 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται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 εγκρίνονται. 10, 11 και 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία, ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 15. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ήταν η 15 αυτή. Τροπολογία 16. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18, 19, 20 μαζί. Συμφωνείτε. 18 με 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 22. Όχι, 21 διορθώνει ο πρόεδρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, αιτιολογική αναφορά. Τροπολογία αριθμός 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροποποιημένη γνωμοδότηση. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε και ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Άλλοι δύο πρέπει να ψηφίσουν ακόμα. Άλλος ένας. Πέρα της φοφορίας. Έκπληξη. 13 υπέρ, 10 ψήφι κατά, καμία αποχή. Καλώς. Ήταν λίγο τσιματσίμα. Συνεχίζουμε και περνάμε στην καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη. Μία βιοοικονομία για την Ευρώπη. Τροπολογία ρυθμός 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ.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 Τροπολογία 6. Σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση από τη τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 μέχρι 14 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Επί της τροποποιηθήσης γνωμοδοτήσεως υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία επί του συνόλου. Πέρας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Συγχαρητήρια στην εξαίρετη εισηγήτριά μας, την κυρία Λέβιν. Περνάμε τώρα στη ψηφοφορία της εκθέσεως για την φιλοκτονία λεστήσεις γυναίκες σε τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 η οποία ζητά ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές. Δεν γνωρίζω, λέει η Πρόεδρος. Oui, c'est l'amendement 2, c'est split c'est Λοιπόν, συγγνώμη, θα ξαναρχίσουμε. Τροπολογία 2 ε, ψηφοφορία τα τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απερίφθη. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Τροπολογία 3. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Ε, θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ωραία. Επί της τροπολογίας 6. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επαλήθευσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. Προφορική τροπολογία υπερθμών 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14, υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροποποιηθεί σε γνωμοδότηση υπέρ. Κατά. Ποιος απέχει ε, εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επαλήθευσης. Le vote est ψηφοφορίας. 21 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στην κυρία Κρετού, η οποία ανταποκρίθηκε σε αυτό το τόσο ε, σύντομο διάστημα, χρονοδιάγραμμα που της δώσαμε. Πολύ ωραία. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας το καρτελάκι της ψηφοφορίας για την επόμενη φορά.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 We have three minutes of suspension. Τρία λεπτά διακόπτουμε. Τρία λεπτά. Περνάμε στο σημείο 23 της ημερήσιας διάταξης τώρα, που αναφέρεται στις θεσμικές πτυχές της, της συνοχής της, των πολιτικών μας υπέρ της ανάπτυξης. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων για αυτό το σημαντικό θέμα με την κοινωνία των πολιτών που εκπροσωπείται εδώ από την Concord. Θα το γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πάρα πολλούς μηχανισμούς και θεσμούς που διευκολύνουν την τήρηση και τον έλεγχο των υποχρεώσεών μας σε σχέση με την συνοχή των πολιτικών μας υπέρ της ανάπτυξης. Ιδιαίτερα έχουμε το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε το άρθρο 12 επίσης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης Κοτονού. Έχουμε τις διάφορες ρήτρες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα μέτρα διασφάλισης, όπως επίσης και μελέτες αντικτύπου. Και παρά την πρόοδο που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθεί να υπάρχει χάσμα ανάμεσα στις προθέσεις και την πραγματικότητα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι όπως αυτές τη ζουν ε, επιτόπου οι άνθρωποι που πλήττονται από την ένδια στις υπανάπτυξη χώρες. Γι' αυτό και πρέπει να ενισχυθούν οι δυνατότητες και οι μηχανισμοί που διαθέτουμε έτσι ώστε να εφαρμόζονται οι υποχρώσεις μας επιτόπου και όντως να υπάρχει συνοχή στις πολιτικές μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επ' αυτού έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Τόσο το Συμβούλιο, το Συμβούλιο όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λογοδοτούν για την εκτέλεση των ε, υποχρεώσεων που έχουν αναλυφθεί στον τομέα αυτό μετά από τις ακροάσεις που είχαμε με τους αρμόδιους επιτρόπους και αναφέρονται μεταξύ άλλων και στη Συμφωνία Κοτονού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν με την κοινωνία των πολιτών και με τις τοπικές αρχές μπορεί να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων ώστε να υπάρχει συνοχή στις πολιτικές μας υπέρ της ανάπτυξης μετά από διαβούλευση και δημοκρατικό διάλογο και στις υπονάπτυξη χώρες αλλά και στις αναπτυγμένες χώρες. Η σημερινή ανταλλαγή απόψεων έχει ως ε, στόχο ο, να ενημερωθεί παρετέρω ο κύριος Γκέρεντ, που είναι ο μόνιμος εισηγητής μας για τις πολιτικές μας στον τομέα της ανάπτυξης. Εννοείται ότι στις συζητήσεις μας προσκαλούμε και εκπροσώπους της Κοντκόρ, που είναι η πλατφόρμα η ευρωπαϊκή των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων για την ανάπτυξη. Είναι η κυρία Λόρα Σάλιβαν από την Action Aid, εκ μέρους της Concord παρεμβαίνει σήμερα εδώ. Καλώς ήρθατε. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκέρενς, που είναι ο μόνιμος εκπρόσωπός μας για την ε, πολιτική συνοχή των πολιτικών μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος για δύο λόγους. Πρώτον, εσείς θέσατε το πλαίσιο της σημερινής συζήτησης. Δεύτερον, η παρουσία της Concord εδώ, με, τη συμμετοχή, με συμμετοχή βέβαια πολύ ενεργό στη συζήτησή μας, εγγράφεται στα πλαίσια τις επιθυμίες τους να παρέμβουν στον διάλογο για την συνοχή των πολιτικών μας. Ήταν κάτι που θέλαμε να το είχαμε κάνει και στη συνάντησή μας με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Δυστυχώς δεν προλάβαμε. Γι' αυτό και αναβλήθηκε. Γι' αυτό και θα ήθελα να πάρει το λόγο η Κονκόρντ ευθύ αμέσω. Να μας πούνε με κάθε ειλικρίνεια ότι έχουν να πούν. Έπειτα, μια που προβλέπουμε, δεν έχει αποφασιστεί βέβαια αυτό ακόμα, ένα εργαστήριο για την συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών μέσα στους επόμενους μήνες, θα ήθελα να μας προτείνει ένα θέμα η Concord ακριβώς για αυτό το εργαστήριο και για να μπορέσουν έτσι να συμμετάσχουν και πιο ανεργά και οι ίδιοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Λόρα Σάλιβαν ε, και εκπροσωπώ την Active International εδώ στο, στις Βρυξέλλες, αλλά είμαστε μέλος της Concord και εργαζόμαστε πάνω στην ε, πολιτική συνοχή, στην ε, αναπτυξιακή συνεργασία. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο σήμερα να μπορέσουμε να μιλήσουμε πριν την κυρία Άστον εδώ σήμερα για να, εμπνεύσουμε, να σας εμπνεύσουμε να θέσετε ερωτήσεις προς την Καθρινά Άστον ε, αργότερα σήμερα. Σήμερα μπήκα στο Google και έψαξα το PCD και τι ε, ε, είδα, Point Cloud Data, το οποίο προφανώς είναι κάποιο είδος ε, ε, αρχείου. Μετά είχαμε Perfume Cosmetics Designs και μετά είχαμε Pussycat Dolls και διάφορα άλλα τέτοια. Ε, ε αυτό που βλέπετε τώρα στη Ροθόνη το είδαμε πολύ μετά. Ε, και δυστυχώς όταν μιλάμε για την πολιτική συνοχή για την ανάπτυξη, αυτό δύο αντιδράσεις συναντάει στους ανθρώπους. Ή μπερδεύονται τελείως ή τους παίρνει ο ύπνος. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε τον κόσμο να καταλάβει περί τίνος μιλάμε όταν μιλάμε για την πολιτική συνοχή στην ανάπτυξη. Είναι ένα θέμα κοινωνικής ε, δικαιοσύνης, δικαιωμάτων, ε, δικαιοσύνης και να μην δίνουμε κάτι με το ένα χέρι που τους το παίρνουμε με το άλλο χέρι. Να τους το θυμίσουμε λοιπόν. Το PCD λοιπόν ε, είναι όχι μόνο τεχνικό θέμα, είναι και πρέπει να είναι πολιτικό θέμα και θα πρέπει εκεί να ξεκινάει. Αυτός λοιπόν είναι άλλος ένας λόγος ε, που χαιρόμαστε που θα μιλήσετε σήμερα με την Καθρίνα Άστον και μπορείτε να θίξετε το θέμα. Οι μηχανισμοί είναι πολύ σημαντικοί για να ε, γίνει η πολιτική βούληση πραγματικές αλλαγές. Γιατί λοιπόν χρειαζόμαστε μηχανισμούς. Καταρχήν, ε, η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Δεύτερον, ε, για να διαπιστώνουμε πότε πραγματικά ε, συμβαίνει και ε, τρίτον να έχουμε δυνατότητα διόρθωσης. Να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε και στους τρεις αυτούς τομείς. Όσον αφορά την πρόληψη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε πολλές εκ των προτέρων και εκ των υστέρων μελέτες αντικτύπου. Θα γνωρίζετε ότι αυτό είναι υποχρεωτικό για πάρα πολλές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για όλες τις μεγάλες η Concord στην Δανία έκανε μια μελέτη που ήταν πολύ δύσκολη και πήρε πολύ χρόνο, αλλά διαπιστώσαν ότι από το διάστημα 2009 μέχρι 2011 μόνο 7 από τις μελέτες αντικτύπου εξέταζαν το θέμα τη ε, της ανάπτυξης. Εμείς αναρωτιόμαστε λοιπόν γιατί, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί δεν μπορούμε με ούτε εκ των προτέρων να έχουμε μελέτες αντικτύπου που να δείχνουν αν υπάρχει αντίκτυπος. Είναι ε, πρόβλημα έλλειψης πολιτικής βούλησης. Ξέρουμε ότι τον ε, περασμένο Μάιο υπεγράφησαν ε, συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ε, αλλά εάν δεν έχουμε καλές ε, μελέτες αντικτύπου, πώς θα το κάνουμε αυτό. Δεύτερον, έχουμε έλλειψη προσωπικού. Οι άνθρωποι που εκπονούν αυτές τις μελέτες που ξέρουν πώς να αναλύουν θέματα ανάπτυξης. Υπάρχει τρόπος να βρούμε ανθρώπους από τις αντιπροσωπείς που μας βοηθήσουν ή απλά υπάρχει έλλειψη ευαισθητοποίησης. Ξέρουμε ότι το θέμα αυτό δεν αναφέρεται ρητά στις κατευθυντήρες γραμμές ε, για το πώς πρέπει να εκπονούνται οι ε, μελέτες αντικτύπου. Υπάρχουν κατευθυντήρες γραμμές ε, που λένε ότι πρέπει να κοιτάει κανείς τις πτυχές της ανάπτυξης, αλλά όχι συγκεκριμένα την πολιτική, την πολιτική συνοχή. Επίσης, όταν το PCD δεν πάει καλά, και έχουμε παραβίαση των δικαιωμάτων. Σήμερα το πρωί μιλήσατε για τα βιοκαύσιμα. Έχουμε ένα ε, παράδειγμα του φετινού Μαρτίου, όπου η Γενική Διεύθυνση Περιενέργειας εκπώνησε μία έκθεση ως μέρος των υποχρεώσεων της από τη σχετική οδηγία να εξετάσει τα δικαιώματα γης, ε, την διαθεσιμότητα τροφίμων ε, και άλλες ε, πτυχές που, σχεδια... που σχετίζονται με την πολιτική ανανεώσιμων πηγών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει λοιπόν στόχος ποσοστού 10% μέχρι το 2020 ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δεν έχουμε αρκετή γη για να το πετύχουμε αυτό, γι' αυτό προσφεύγουμε στον αναπτυσσόμενο αναπτυσσόμενο κόσμο. Ε, ουσιαστικά στερούμε από τον κόσμο την τροφή του και αυτό επίσης επηρεάζει και τα εργασιακά δικαιώματα των ανθρώπων. Στη συγκεκριμένη μελέτη δεν είχαμε μελέτη επιτόπου. Ε, σε αντίθεση με αυτό που έκανε πρόσφατα η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξη, ε, που είχε δύο μελέτε από τη Σενεγάλη και την Τανζανία. Η Γενική Διεύθυνση Ενέργεια βασίστηκε σε μελέτε τη ΕΚΟΦΗΣ και χρησιμοποιεί μόνο μία πηγή ε, ακαδημαϊκή ε, δεν εξετάζει πολλές μελέτες μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων. Εξετάζει μόνο το διάστημα μέχρι το 2010 ενώ η οδηγία ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργεια υιοθετήθηκε ένα χρόνο πριν. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να αξιολογήσει κανεί τον αντίκτυπο. Επίση, δεν εξετάζει, υποτιμάει μάλλον τι επιπτώσει των τιμών των τροφίμων. Ε, τρίτον, έχουμε το θέμα ε, αντιμετώπισης του αντικτύπου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει κάποιο πραγματικό σύστημα που να βοηθάει τις ε, κοινότητες ε, που πλήττονται να ε, προωθήσουν θέματα PCD. Δηλαδή, εάν μια κοινότητα στην Κένια χάσει τη γη της επειδή κάποια Ιταλική εταιρεία θέλει να εξάγει βιοκαύσιμα στην Ευρώπη, πού μπορούν να προσφύγουν. Αυτή τη στιγμή πουθενά δεν μπορούν να προσφύγουν. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να δούμε τι ακριβώς γίνεται επί τόπου και όχι μόνο να έχουμε τις γνώσεις αυτές, αλλά να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πραγματική ευκαιρία εδώ πέρα ε, είναι ευκαιρία για τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να ε, συλλέξουν τις πληροφορίες αυτές και να τις στείλουν πίσω στις Βρυξέλλες. Πιστεύουμε ότι χάνουμε μια σημαντική ευκαιρία διότι οι αντιπροσωπείες ζητούν τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας των πολιτών. Μήπως λοιπόν είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της χώρας αυτής. Και ολοκληρώνω. Πρέπει να πιέσουμε τους ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να ε, διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν ε, ε, μηχανισμοί προσφυγής για τους πολίτες, διότι αλλιώς η συνθήκη της Λισαβόνας δεν θα έχει κανένα νόημα. Μία πολύ σύντομη διαφάνεια, ελπίζω να μπορώ, να μπορώ σας τα διανύμω αυτά αργότερα. Πάντως υπάρχει ένα πολύ καλό παράδειγμα από το Δανέζικο Κοινοβούλιο που προσπαθεί να εξετάσει την ε, ε, πολιτική ανάπτυξη. Σε η ε, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μπορεί να συνομιλεί με όλους τους υπουργούς ώστε να έχει, ε, ώστε να έχουν εντολή να ε, μιλήσουν για συγκεκριμένα θέματα συμπεριλαμβανομένου και του PCDPD. Ε, δεν ξέρω ακόμα αν το έχουν χρησιμοποιήσει σε συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλή πρακτική. Και οι δύο τελευταίες ε, διαφάνειες, ποιες είναι οι συστάσεις μας ε, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και προς εσάς ως Επιτροπή Ανάπτυξης. Καταρχήν, πρέπει να επικαλεστούμε την πολιτική βούληση, πρέπει να επιβεβαιώσουμε την πολιτική βούληση σε υψηλότερο επίπεδο. Τι κάνουν οι ηγέτες μας για αυτά, τι κάνει η Καθολίνα Άστον και τι λέει για τα, για τα θέματα αυτά. Το ίδιο ισχύει για τον Παρόσο και τον Επίτροπο Πίμπαλξ. Πρέπει την Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης ε, και το Συμβούλιο να τους ε, επιστήσουμε την προσοχή στα περσινά ε, συμπεράσματα. Πρέπει οι τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής Ε, αλλά ε, αυτή τη στιγμή ε, απλά περιμένουμε επιστολή με κατευθυντήριες γραμμές για όλα αυτά. Εάν περιμένουμε ένα χρόνο μια επιστολή, πόσο χρόνο θα πάρει η πραγματοποίηση όλων αυτών. Πρέπει να απαιτήσουμε να υπάρξει πρόοδος για μηχανισμούς προσφυγής, διότι είναι ο μόνος τρόπος να μπορούμε να έχουμε δικαιοσύνη και όλα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος των συζητήσεων ε, για το πλαίσιο μετά το 2015. Όταν μιλάμε για την ανάπτυξη, δεν μιλάμε μόνο για ε, χρηματοδότηση. Ε, Επίση σημαντικό πρόβλημα, πολύ σημαντικό θέμα είναι να μην βλάπτουμε τις χώρες αυτές. Επίσης, θέλω να μιλήσω μαζί σας για κάποιες από τις προτάσεις που έχετε υποβάλει εσείς και που θα μπορούσαν να προωθηθούν. Να ενισχυθεί ο ρόλος του μόνιμου εισηγητή για το PCD μετά το 2014. Πιστεύω ότι ο εισηγητής αυτό ε, χρειάζεται προσωπικό και θα πρέπει ε, να ε, συνεχίσει να υπάρχει και στην επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου μετά το 2014. Σύμφωνο με αυτούς που λένε ότι είναι κάτι που αφορά όχι μόνο την Επιτροπή Ανάπτυξης αλλά και άλλες επιτροπές. Αυτές λοιπόν οι διεπιτροπικές σχέσεις θα πρέπει να συνεχιστούν. Μίλησα με κάποιον από την Επιτροπή ε, Απασχόλησης. Θα θέλαμε πολύ να ξεκινήσουμε ε, με αυτά τα θέματα, ε, να συζητώνται τα θέματα αυτά και σε άλλες επιτροπές. Χρειαζόμαστε εισηγητές για το PCD και στην κοινή κυροβουλευτική συνέλευση διότι είναι σημαντικό και η πλευρά ΑΚΕ ε, να ασχοληθεί με το PCD. Επίσης, έχετε κάνει ένα πολύ καλό βήμα, αλλά θα πρέπει να ενταθούν οι σχέσεις ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια πάνω στο PCD. Πρέπει επίσης να τεθεί στο θεματολόγιο ε, της μονάδας ε, του Κοινοβουλίου για τις μελέτες αντικτύπου και επίσης θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή στην φετινή ή νομίζω του χρόνου πρόκειται να γίνει θεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις μελέτε αντικτύπου που δεν αναφέρουν καθόλου το PCD. Ε, αυτές λοιπόν είναι τεχνικές συστάσεις, ε, πιστεύουμε όμως ότι είναι κάποιε που μπορείτε να προωθήσετε. Αυτά αυτή τη στιγμή. Ε, πολύ ευχαριστώ, θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. <coughs> Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Όποιος ε, θέλει από τους παριστάμενους βουλευτές ε, μπορεί να ζητήσει και να πάρει το λόγο έχοντας ακούσει την παρέμβαση της κυρίας Σάλιβαν ε, η οποία με μεγάλο πάθος και ενεργητικότητα έκανε την παρουσίασή της και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριος Γκέρενσε θα ήθελε ενθερμό να αντιδράσω στα όσα ακούσαμε μόλις. Και θα συμφωνήσω με το σχόλιο που κάνατε. Ήταν ε, πραγματικά ε, ε, και μεγάλη χαρά να σας ακούσει κανείς, γιατί είσαστε και παθιασμένοι και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Πριν έρθω εδώ είχαμε και μία ανταλλαγή απόψε με τον Επίτροπο Πίμπαλτσα στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου και η ερώτησή μου προς αυτόν αφορούσε ακριβώς το είδος του εγγράφου που θα μας υποβάλει η Κομισιόν τον Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, το αργότερο τον Οκτώβριο. Εμείς θα επιθυμούσαμε, εγώ τουλάχιστον, ε, εάν μπορώ να θεωρήσω ότι είμαι εκφραστής ε, της ε, απόψεως της Επιτροπής μας, Εάν λοιπόν μπορώ να το κάνω αυτό, θα έλεγα ότι θα προτιμούσαμε το καθεστώς ε, μιας ανακοίνωσης και όχι το καθεστώς ε, μιας απλής έκθεσης. Θεωρούμε ότι μέσω της ανακοίνωσης αποδίδεται και σημασία στο περιεχόμενο της ε, ανακοίνωσης και ταυτόχρονα και στη δικιά μας τη δουλειά. Δεύτερον, μέχρι τότε θα έχουμε στα πλαίσια της Επιτροπής δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και μια και είναι ένα θέμα που διαρκώς επανέρχεται, επανέρχεται ακριβώς και σε όλες τις ανταλλαγές απόψεων που έχουμε ε, με την ε, Κομισιόν. Και άλλωστε και στην Λεδιάστον θα έχω τη δυνατότητα να υποβάλω το ίδιο ερώτημα. Θα έχουμε και συνάντηση με εξωτερικούς ε, εμπειρογνώμονε στα πλαίσια ενός εργαστηρίου που ενδεχομένως θα διοργανωθεί πριν το καλοκαίρι ή εν πριν τι καλοκαιρινέ διακοπές. Στα πλαίσια αυτού του εργαστηρίου θα ήθελα πραγματικά να είστε κι εσείς ε, παρούσα. Όπως και σήμερα ε, η θεματική ε, απεριστρέφεται γύρω από την μεθοδολογία. Καλό θα ήταν να μας προτείνετε ένα θέμα, αλλά οπωσδήποτε να εκφραστεί και η Concordo, η πλατφόρμα αυτή, επί της μεθοδολογίας που εσείς θα προτιμούσατε να επιλεγεί ε, στα πλαίσια της ε, προσέγγισης, της ακολουθητέας προσέγγισης και νομίζω ότι άλλωστε το ίδιο γίνεται και με τον ε, ΟΣΑ που ήδη στον τομέα της αξιολόγησης έχει κάνει ε, πολύ πρωτοποριακή δουλειά. Είναι το πρώτο θεσμικό όργανο το οποίο ε, προτείνει και προχωράει στην αξιολόγηση των αναπτυξιακών πολιτικών. Και μια και στον ΟΣΑ έχουν ήδη ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση για το θέμα αυτό. Η βοηθός μου Κριστίν ε, πηγαίνει και παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις με το θέμα αυτό του στο ΝΟΣΑ, στο Παρίσι. Θα έχουμε επίσης, διάβασα κάτι τέτοιο, θα έχουμε και την, την επίσκεψη του νέου Προέδρου ε, της ε, Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του Όσα που θα έρθει ενώπιόν μας για να ακριβώς να, αναπτύξει το θέμα αυτό. Και επομένως καταλαβαίνετε ότι είναι μια εργασία η οποία βεβαίως δεν θα σταματήσει με την έκθεση αυτή. Μετά την δημοσίευση της εκθέσεως ή το ελπίζουμε, της ανακοίνωσης της Επιτροπής θα υπάρξει αντίδραση μέσω εκθέσεως, η οποία θα δημοσιευθεί Ιανουάριο-Φεβρουάριο και που θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Και επομένως ε, θα είναι μία έκθεση η οποία θα λαμβάνει υπόψη όλες τις προτάσεις ε, που θα έχουμε ακούσει στον διάλογο που θα έχουμε και με την Κομισιόν αλλά και στο εργαστήριο το οποίο ε, ανέφερα προηγουμένως. Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση εν θερμό. Φαντάζομαι ότι και άλλοι συνάδελφοι μπορούν να μιλήσουν επί του θέματος αυτού. Εγώ να πω μονάχα ότι δεν δεν, ε, δεν είμαι ο πρώτος ο οποίος ασχολήθηκε με την συνοχή αναπτυξιακών πολιτικών. Θεωρώ και εγώ βεβαίως ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά έχουμε ήδη μια συνάδελφο η οποία πρώτη είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό ε, στην έκθεσή της και η ουσία εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά βεβαίως δεν πρέπει, γιατί είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική, να παραβλέψουμε την μεθοδολογία. Ε, επίσης να πω ότι δεν έχουμε πλέον ε, καμία άλλη πρωτοβουλία πέραν ε, αυτής ε, του 2015 που θα ονομαστεί έτος ανάπτυξης ε, και εγώ ορίστηκα εισηγητής ακριβώς για τη συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών και θα είμαι συνέχεια εισηγητής για την, για την Επιτροπή μας. Ο κύριος Γκούσταυσον θα μιλήσω σου ειδικά εάν δεν γνωρίζετε παρελπίδα την γλώσσα αυτή παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Ήταν ξεκάθαρη και πολύ συγκεκριμένη. Ήταν πολύ εύκολο για έναν πολιτικό να καταλάβει τα συμπεράσματα και η παρουσίαση αυτή συμπεριλαμβάνει πολλά σημαντικά στοιχεία Γι' αυτό ε, ε, είναι πολύ δύσκολο να σε ρωτήσω τι θέλεις να κάνουμε, διότι ήσουν πάρα πολύ σαφής. Ε, σε ευχαριστώ που ήρθες και ευχαριστώ και όλες τις οργανώσεις που βοηθούν εμάς τους πολιτικούς. Είναι πολύ σημαντικές οι οργανώσεις αυτές για μας, διότι έχετε γνώσεις στον τομέα αυτών που δεν έχουμε εμείς. Στις οι ανταλλαγές αυτές λοιπόν μαζί μας μας βοηθούν στην εργασία μας ε, μας βοηθούν να κάνουμε πιο συγκεκριμένες ε, κάποιες ιδέες μας. Ε, ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να λάβουμε με email ή με κάποιο άλλο τρόπο αυτή την παρουσίαση PowerPoint. Διότι υπήρχαν πολύ σαφείς ιδέες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο τώρα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Στέγκα τον Πιάσοβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Concord για την πολύ καλή παρουσίαση της ε, με πολλές ε, προτάσεις. Ε, κάποιες από αυτές απευθύνονται και σε εμά. Αναγνωρίζουμε την ε, σημασία της μεθόδους αυτής. Ε, συνεχίζουμε να, τις προσπάθειές μας να βελτιώσουμε ε, την χρησιμότητα των μελετών αντικτύπου για το PCT. Προσπαθούμε να συμπληρώσουμε τα κενά που υπάρχουν στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απτυσιακή βοήθεια και δεν νομίζω ότι είναι μυστικό αυτό. Συνεργαζόμαστε στενά με τον ΩΣΑ και μάλιστα πριν έρθουμε εδώ πέρα. Είχαμε μια πρόσκληση για ε, άλλη μια συνάντηση επιρογνωμόνων ε, στον ΟΣΑ για ε, την παροχή τροφίμων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε βρει ακόμα τη λύση θαύμα που αλλά όλα αυτά θα αποτελέσουν στοιχεία της έκθεσής μας. Αυτή τη στιγμή ε, είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε την επιστολή μας προς τις αντιπροσωπείες, αλλά είναι στα σκαριά η δουλειά αυτή. Ε, παρακαλούμε υπομονή, θέλει λίγο περισσότερο χρόνο όταν στέλνει επιστολή, επιστολή η Επιτροπή και όχι ε, ένα πρόσωπο. Θέλουμε πάρα πολύ να συμπεριλάβουμε τις ε, εργασίες PCD στις υπόλοιπες εργασίες μας οι αντιπροσωπείες μάλλον θέλουν να το κάνουν αυτό και δεν θέλουμε να προσθέσουμε να τους δώσουμε ακόμα περισσότερη δουλειά. Προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε το υλικό που λαμβάνουμε από τις αντιπροσωπείες. Ε, δεν πρόκειται λοιπόν απλά για μία επιστολή. Ε, δεν ε, χρειάζεται να, να κάνουμε συζήτηση. Ήδη ακούσατε τον Επιτροπό μας. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα όσα είπε ήδη σήμερα. Ευχαριστώ. Merci Σας ευχαριστούμε. Τώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ο κύριος Φίλιξ Φερνάντισον να μας μιλήσει, να μας παρουσιάσει την άποψη της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης όσον αφορά τη συνοχή των αναπτυξιακών μας πολιτικών. Ευχαριστώ κύριε Ζολή και ευχαριστώ τη Λόρα για την παρουσίασή της. Θα συμφωνήσω και εγώ με τον κύριο Γκέρενς για το ότι την παρουσίασε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Και όλοι συμμεριζόμαστε αυτό τον ενθουσιασμό, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε για να πετύχουμε τους στόχους. Ιδιαίτερα οι αντιπροσωπείες, οι οποίες δεν έχουν αρκετό προσωπικό. Αλλά επιβεβαιώνω αυτό που λέει και η Κομισιόν, ότι δηλαδή συνεργαζόμαστε με τη Γενική Διεύθυνση ΑΦΚΟ για να δίνουμε οδηγίες στις αντιπροσωπείες όσον αφορά τη συνοχή της αναπτυξιακής βοήθειας. Πώς θα έχει συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και πώς θα καταλήγει σε καλύτερες εκθέσεις. Δεν είναι βέβαια εύκολη δουλειά. Εννοείται. Το δουλεύουμε πάντως και όταν έχουμε κάτι έτοιμο θα επανέλθουμε. Πρόεδρος, Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει πάλι εκπρόσωπος της κοινωνίας των πολιτών. Η κυρία Λόρα Σάλιβαν. Ευχαριστώ. Θέλω να δώσω κάποιες απαντήσεις. Να πω στον κύριο Γκέρενς πρώτα απ' όλα ότι ευχαρίστως να έρθουμε στο εργαστήριο αυτό που λέτε ότι θα οργανωθεί. Μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ θεματικά, πιέζοντας για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και στους μηχανισμούς. Δεν μπορώ να σας πω από τώρα ποιο θα είναι το θέμα, αλλά να ξέρετε ότι εμείς ετοιμάζουμε την έκθεσή μας και θα είναι έτοιμη την εποχή του εργαστηρίου και που θα λέει σε ποιου θεματικούς τομείς δεν έχουμε πετύχει τη συνοχή. Θα σας κρατώ ενήμερο πάντως. Σίγουρα δεχόμαστε την πρόσκληση. Όσον αφορά τώρα τόσο ακούσαμε από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ειλικρινά, συνεργαζόμαστε πολύ καλά και με τις δύο αυτές μονάδες. Ξέρω ότι παίρνουν τη δουλειά αυτή πολύ στα σοβαρά. Περιμένουμε τις κατευθυντήριες γραμμές για τις αντιπροσωπείες, αλλά θα ήθελα να ενθαρρύνω και την Επιτροπή σας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να δει και να παρακολουθήσει τι θα γίνει μετά. Γιατί καλά, φτάνει η πληροφορία στις αντιπροσωπείες. Μετά όμως τι θα γίνει. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος της βελτίωσης. Τι θα γίνει στις Βρυξέλλες. Οπότε ευχαριστώ πολύ. Ευχαρίστως να συνεχίσουμε το διάλογο μαζί σας. Και αν θέλετε πιο συγκεκριμένα παραδείγματα, ευχαρίστως να σας τα δώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γκέρενς για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Ε, η εκπρόσωπος του Concord κατέληξε πολύ καλά σε συμπεράσματα, αλλά εγώ θα προσθέσω κάτι που ξέχασα πριν. Πρέπει να συμφωνήσουμε για το ποια είναι η περίμετρος της αξιολόγησης της συνοχής αναπτυξιακής μας πολιτικής. Θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι ο αντίκτυπο τη πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών επί τη ανάπτυξη. Δεν είμαστε όμως οι μόνοι που δρούμε, που σημαίνει ότι μια καλή δικιά μας δράση μπορεί να χαλάει από την κακή δράση κάποιου άλλου φορέα. Έχουμε λοιπόν την τάση να μιλάμε αρνητικά για οτιδήποτε έχει να κάνει με την αναπτυξιακή συνεργασία. Δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να υπάρχει διαφοροποίηση στην αξιολόγηση. Γι' αυτό και περιμένω περισσότερα στοιχεία από αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση στην έκθεσή του. Γιατί είναι ζωτική σημασία. Για έναν πολύ απλό λόγο. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός φορέας όταν πρόκειται για αναπτυξιακή βοήθεια, η ευθύνη της, όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη. Πρέπει λοιπόν να αξιολογούμε πολύ ορθά τον αντίκτυπο της πολιτικής της. Είναι πολύ ιδιαίτερη η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό φαίνεται στις μεγάλες συζητήσεις που έχουμε. Για παράδειγμα, όταν συζητήσαμε τους στόχους της χιλιετίας για, τους, για το μετά του 2015. Πάντως, μόνο θετικά σχόλια έχω για τόσα μας είπε η Concord, η κυρία Σάλιβαν πιο συγκεκριμένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την αντιπροσωπεία που έφτασε εδώ για να παρακολουθήσει τις εργασίες της Επιτροπής μας. Είναι πολιτικοί ηγέτες από το Σουδάν οι οποίοι έρχονται στα πλαίσια ε, της δράσης μας για την προώθηση του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Καλώς ήρθατε. Σε λίγο θα έχουμε εδώ την είπα το εκπρόσωπο, την κυρία Άστον μαζί μας. Συνεπώς, λίγε το σημείο αυτό για τη συνοχή της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Και θέλω να διαβεβαιώσω την κοινωνία των πολιτών ότι το σημείο αυτό δεν θα εξαφανιστεί ποτέ από την ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Ωραία. Ολοκληρώσαμε την ημερήσια διάταξη μέχρι την άφηξη της κυρίας Άστον. Στις 5.30 την περιμένουμε. Διακόπτουμε συνεπώς μέχρι τις 17 και 28. Στις 17 και 28 παρακαλώ να είσαστε εδώ. Ευχαριστώ.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 Ας καθίσουμε αγαπητοί συνάδελφοι έτσι ώστε να υποδαχθούμε την ύπατη εκπρόσωπο.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 Euh, Πρόεδρος, με μεγάλη χαρά υποδέχομαι την ε, Βαρόνια Άστον, ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τις ε, εξωτερικές υποθέσεις και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με την ευκαιρία της ετήσιας επίσκεψής της στην Επιτροπή μας. Κυρία Έστον, Πάντα με μεγάλη χαρά ε, ε, βλέπουμε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας και να έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Οι υπηρεσίες σας ζουν, ε, παίζουν πράγματι έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην, πολιτική, στην αναπτυξιακή πολιτική, ιδιαίτερος δε όσον αφορά τον προγραμματισμό των δράσεων των επιχειρήσεων ε, μέσα στα πλαίσια του εργαλείου για την συνεργασία και την ανάπτυξη, καθώς επίσης και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Αυτό ε, μας ενδιαφέρει και ενδιαφέρει ιδιαίτερο στην Επιτροπή μας, ε, γιατί συμμερίζεται το σχέδιο της υλοποίησης ε, του μελλοντικού προγράμματος σε ορισμένες ε, χώρες από κοινού με τα κράτη-μέλη. Η, πρόταση, η επίσκεψή σας πραγματικά έρχεται την κατάλληλη στιγμή ε, γιατί η συνάντηση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων οπου αφορά ανεπτυξιακά θέματα έλαβε χώρα σήμερα το πρωί υπό την Προεδρία σας κυρία Άστον και επομένως θα έχετε τη δυνατότητα να μας πείτε έχοντας η ίδια ακούσει τις τις ε, ε, τι αποκομίσατε από αυτές. Οι αρμόδιοι Υπουργοί Ανάπτυξης αναφέρθηκαν ε, σε πολλά θέματα πολύ σημαντικά, τα οποία είναι ιδιαίτερος προσφυλή στην Επιτροπή μας. Θα σας ακούσουμε λοιπόν με πολύ μεγάλη προσοχή και χωρίς καθόλου να μακρηγορήσω, θα σας δώσω αμέσως το λόγο κυρία Άστονα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης και που σας ξαναβλέπω κυρία Ζολή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλη τη δουλειά που έχει κάνει. Έχουμε εδώ παρόντες και νέους ηγέτες από το Σουδάν. Ε, σας χαιρετίζω και σας λέω ότι είναι μεγάλη μας τιμή και θεωρούμε πολύ σημαντική την παρουσία σας εδώ. Ελπίζουμε ότι ε, θα κερδίσετε, θα αποκομίσετε πολλά από αυτήν την επίσκεψη. Ε, θα σας δώσω κάποιες πληροφορίες ε, σχετικά με τα όσα έλαβαν χώρα σήμερα το πρωί. Όπως υποσχέθηκα και σε εσά εδώ αλλά και στα κράτη-μέλη, θα έχουμε πλέον μία μέρα αφιερωμένη στα θέματα ανάπτυξης Σήμερα συζητήσαμε και για το τι θα γίνει μετά το 2015, καθώς επίσης και τι θα γίνει όσον αφορά ε, την ε, ατζέντα για, την, ε, για τις αλλαγές που θα λάβουν χώρα μετά. Νομίζω ότι προηγουμένως είχατε και τον Επίτροπο Πίτμπολης εδώ και σας ανέφερε πολλά θέματα και ε, βεβαίως για το 2015 και μετά έχουμε πολλά θέματα και το Αφγανιστάν και τη Μιανμάρ. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα για το 2015. Ξέρετε ότι το πιο πιεστικό είναι ε, το τι ε, γίνεται με τους αναπτυξιακούς στόχους και τι θα γίνει με την παρακολούθηση των προγραμμάτων για τα επόμενα 20 χρόνια. Τι θα γίνει όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. του έχουμε προετοιμάσει τους στόχους αυτούς, θέλουμε να δούμε τι θα γίνει μετά. Ε, θέλουμε ε, μια, ένα συνολικό πλαίσιο να οικοδομήσουμε για την περίοδο του 2015 ε, έτσι ώστε να ε, έχουμε ένα ε, και μόνο πλαίσιο με πολλές ιεραρχημένες προτεραιότητες. Αυτό βεβαίως ε, δεν είναι εύκολο και δεν είναι καθόλου εύκολο και να διατηρήσουμε και την συνοχή όλων αυτών των πολιτικών. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς αλλά και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για τα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα. Είπαμε ότι ε, τα επιτεύγματά μας και οι προσπάθειές μας μάλλον θα πρέπει να είναι συνολικές και καθολικές. Να αφορούν όλες τις χώρες συμπεριλαμβανομένων και των αναδειωμένων οικονομικών. Ε, είπαμε ότι η δημοκρατική διακυβέρνηση και ο σεβασμός ε, των δημοκρατικών κανόνων και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι από τις εκ των ουκάνευ για την αηφόρο ανάπτυξη. Δεν θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι ε, συμμερίζονται την ε, ίδια άποψη, αλλά η στήριξη του Κοινοβουλίου επ' αυτού θα είναι πάρα πολύ σημαντική και βεβαίως ε, περιμένουμε αδημονία την έκθεση του κ. Κάσμαράκα. Ένα άλλο ε, θέμα είναι η ε, ε, ατζέντα της αλλαγής και το χρηματοδοτικό εργαλείο 15, για την περίοδο 2015-2020. Προσωπικά πιστεύω ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουν ακριβώς το ίδιο βάρος σε αυτήν την διαπραγμάτευση. Όπως γνωρίζετε, ο στόχος είναι να έχουμε σαφή αναπτυξιακή πολιτική ε, με συνέχεια και συνέπεια. Να μεγιστοποιήσουμε την επιρροή που έχουμε και τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει αυτή. Και βεβαίως να στηρίξουμε την ιδέα ότι δεν μπορεί να υπάρξει αηφόρος ανάπτυξη εάν δεν υπάρχει και ειρήνη ε, και αν δεν υπάρχει και ασφάλεια. Ε, προχωρήσαμε με γρηγορότερο ρυθμό, προοδεύσαμε περισσότερο από όσο ε, νομίζαμε. Και μέχρι το 2014 θα έχουμε 20 ε, συνομιλήτριες χώρες, οι οποίες σύντομα θα φτάσουν τον αριθμό των 40. Είμαι ευγνώμων προς τα κράτη-μέλη που στήριξαν μέσω των πρωτευουσών τους και μέσω των ε, ε, πρεσβειών τους επιτόπου τα προγράμματα αυτά, ας πούμε, στην Αιθιοπία όπου ε, η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στενά συνεργάστηκε με, τους 13, με τις 13 εκπροσωπούμενες χώρες μέσω των πρεσβειών. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω εδώ τον Σαντί Μασάλ ε, ο οποίος ε, απεβίωσε πριν από μερικές μέρες, ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, και ήταν πραγματικά υπερασπιστής όλης αυτής της εργασίας επιτόπου στην Αφρική. Θα ήθελα να εκφράσω την θλίψη μου και τα συλληπιτήριά μου προς την οικογένειά του, η κυρία του θα γίνει σε μερικές μέρες. Ε, είχατε και εσείς εδώ στην Επιτροπή ε, μια κοινή συνάντηση με εθνικά κοινοβούλια έτσι ώστε να συζητήσετε την δυνατότητα μεικτών συνεργασιών. Αυτή ακριβώς είναι ε, η προς... αυτός είναι ο δρόμος που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, υπουργούς που παραμένουν ε, πιστοί και δεσμευμένοι στο θέμα της ε, ανάπτυξης και που προσπαθούν να αντλήσουν χρηματοδότηση που δεν είναι καθόλου που δεν είναι καθόλου ε, εύκολο πράγμα σε αυτούς τους ε, χαλεπούς ε, καιρούς. Ξέρουμε, διαβάσαμε και την δήλωση του ΟΣΑ ότι παρά την κρίση η Ευρώπη παραμένει ο μεγαλύτερος χορηγός και δωρητής. Εγώ ζητώ τακτικά και διαρκώς από τους Υπουργούς να παραμένουν προσδεδεμένοι σε αυτές τις δεσμεύσεις ο ρόλος μας, η ηγεσία μας, ο ηγετικός μας ρόλος δεν πρέπει να αμφισβητείται και πρέπει να είμαστε ακόμα πιο αξιόπιστοι, να προσπαθούμε και να μπορούμε να κινητοποιήσουμε χρηματοδότηση από, πολλές, ε, ε, από πολλούς και να χρησιμοποιούμε όλες τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν καταλήτη των διαφόρων διεργασιών. Ε, θα επανέλθουμε βεβαίω στο θέμα αυτό το Σεπτέμβριο με την ανακοίνωση για την ανάπτυξη. Ε, λοιπόν, τώρα Αφγανιστάν και Βυρμανία, Μιανμάρ. Είμαστε πάντα ιδιαίτερα στρατευμένοι στο θέμα του ε, Αφγανιστάν και στους επόμενους μήνες θα ξεκινήσει αυτό που κάποιος θα μπορούσε να ονομάσει τελική φάση της μετάβασης, δηλαδή να ξεκινήσει πλέον η πραγματική ανάπτυξη. Ε, έχουμε ζητήσει τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν την ε, βοήθεια των 200 εκατομμυρίων τουλάχιστον ε, ανά έτος, αλλά βεβαίως θα πρέπει να υλοποιηθεί και το δεκαετές πρόγραμμα στήριξης του Αφγανιστάν. Θα πρέπει τώρα να ξεκινήσει η φάση ε, της ανασυγκρότησης, της θεσμικής ανασυγκρότησης της χώρας και ο Πρόεδρος Αλίας ε, άλλωστε αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Πρέπει στο Αφγανιστάν να διασφαλίσουμε την συνέχεια ε, να δουλέψουμε για το χώρο της δικαιοσύνης, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα. Για την Βερμανία Μιανμάρ ε, έχει ξεκινήσει η μεταβατική περίοδος, αλλά γνωρίζετε όλοι, όπως και εμείς, ε, ότι πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί η ένδια ε, και θα πρέπει να αποκατασταθεί η ηρεμία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αλλαγή των νοοτροπιών και των θέσεων στάσεων δεν θα είναι καθόλου εύκολο να πρέπει να προσπαθήσουμε. Έχουμε αυξήσει την ε, βοήθεια για το 12-13 στα 150 ε, εκατομμύρια. Και ε, θα ηγηθώ τον Νοέμβρη μια task force η οποία θα προσπαθήσει να κινητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους τους ε, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ε, τους πολιτικούς, ε, αλλά και ομάδες επιχειρηματιών κτλ. Ε, κυρία Ζολή, θα μπορούσα να μιλάω επί ώρες για πάρα πολλά θέματα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει εσείς να έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε ερωτήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μίτσελ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Ναρονιάστον. Καλώς ήρθατε. Σίγουρα υπάρχουν πολλά θέματα που θέλουμε να καλύψουμε, αλλά πρώτα απ' όλα να σας πω ότι πολύ χαίρομαι για την ημέρα και την ανάπτυξη που μας αναφέρατε. Διότι είναι τραγικό το ότι μειώνεται το ποσό που πάει στην ανάπτυξη και σε σχέση με το ΑΕΠ. Συρία, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα όπλα στη Συρία. Είναι θέμα κρατών μελών, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα κάνει. Βλέπουμε ότι η Επιτροπή τώρα δραστηριοποιείται περισσότερο στις χώρες που παίρνουν αναπτυξιακή βοήθεια και θέλουμε για κάθε ευρώ που δίνουμε να υπάρχει μόχλευση και να είναι μεγαλύτερο το κέρδος στην ανάπτυξη. Ξέρουμε ας πούμε ότι η Κίνα το φροντίζει αυτό για τα 3,5 δις που δίνει, θέλει να υπάρχει τέτοιο αντίκρισμα. Προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, μα ακριβώς γι' αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή που έχουμε μπροστά μας. Το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω είναι για την φιλοκτονία σε βάρος των γυναικών. Σήμερα είχαμε μια γνωμοδότηση, η Επιτροπή μας, για μια έκθεση που ετοιμάζει η Επιτροπή Γυναικών για αυτό το θέμα. 200 εκατομμύρια γυναίκες λείπουν στο παγκόσμιο πληθυσμό σύμφωνα με τα δεδομένα του ΟΙΕ. Στην Κίνα το 1982 ήταν 100-100 αγόρια κορίτσια. Σήμερα είναι 120 αγόρια και 100 κορίτσια στην Κίνα. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση η Κίνα. Αφήνουν τα κορίτσια, τα μωρά, να πεθαίνουν. Υπάρχει στην έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου. Κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει εμείς να ηγηθούμε μιας εκστρατείας κατά του φαινομένου αυτού. Ο κύριος Κόρτες Λάστρα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Βαρονιάστον, που ήρθατε. Ξέρουμε ότι εσείς προσωπικά στηρίζετε την αναπτυξιακή βοήθεια και από πριν που ήσασταν αρμόδια για το εμπόριο. Σε όλα σας τα ταξίδια και στις συναντήσεις σας υψηλού επίπεδου, ε, πάντα φροντίζετε για να είναι αποτελεσματική αναπτυξιακή μας βοήθεια. Υπάρχει και το έγγραφο το οποίο αναλύει την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας σας τα τελευταία τρία χρόνια. Ξέρουμε ότι το έργο υπάρχει και ας μην προβάλλεται όσο θα θέλαμε, ο αντίκτυπος όμως υπάρχει και τον εκτιμάνε όσοι υποφελούνται από αυτόν. Πρέπει να υπάρχει βεβαίως ε, συνεργασία ανάμεσα στην Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις υπηρεσίες σας. Και οι δύο πλευρές πρέπει όμως να κάνουν περισσότερη προσπάθεια για να καταλήγουν από κοινού σε αξιολογήσεις και από κοινού σε στρατηγικές. Και εδώ έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα. Τώρα έρχομαι στις ερωτήσεις μου, κυρία Άστον. Πρώτον, Ξέρετε ότι η συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών είναι κάτι στο οποίο προχωράμε πολύ αργά. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσετε εσείς τη συνοχή των αναπτυξιακών μας πολιτικών. Γιατί εμεί πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω. Και δεύτερον, παρατηρούμε ένα πραγματικό πρόβλημα με τα ατομικά προγράμματα, τα εγκάρσια, έχουμε το εμπόριο από τη μία την ανάπτυξη, από την άλλη η υπηρεσία σας τι μπορεί να κάνει για να βελτιώσει την κατάσταση σε αυτό το τομέα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκέρενς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ χαιρετίζω εδώ την Lady Άστον και τους συνεργάτες της. Έχουμε εμπειρία από συνεργασία. Στην αρχή ήταν δύσκολο, αλλά τα πράγματα ομολογώ με απόλυτη αντικειμενικότητα ότι έχουν βελτιωθεί. Δεν λέω ότι είναι όλα τέλεια και θα σας εξηγήσω γιατί, αλλά έχουν βελτιωθεί. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα παγκόσμιο οδέρο. Ωραία, συμφωνούμε. Είμαστε οι πρώτοι στην αναπτυξιακή βοήθεια. Ναι, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Επίσης είμαστε αξιόπιστος εταίρος, αν και μπαίνουμε σε ένα χώρο που δεν πρέπει να υποτιμάμε. Συνεπώς πρέπει να αναρωτηθούμε ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίω. Στρατιωτικά εννοείται ότι δεν είναι υπέρ μας τα πράγματα. Στρατηγική, οικονομικά έχουμε βάρος ακόμα, αν και χάνουμε κάπως σε σχέση με άλλους εταίρους αναδιόμενους. Εκεί που μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τη διαφορά και γι' αυτό και γινόμαστε έξαλλοι, γιατί δεν υπάρχει αρκετή προβολή σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι ότι έχουμε το know-how, αλλά δεν το ξέρουν οι άλλοι. Έχουμε ένα πρόβλημα προβολής του έργου μας. Αυτό που είναι ζωτική σημασίας είναι ότι συνεισφέρουμε σημαντικά Μπορούμε να είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητές σε και βοήθεια και πρέπει να παραμείνουμε πρώτοι και να φροντίσουμε οι 28 εταίροι να συνεργάζονται μεταξύ τους. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται περισσότερη συνοχή. Το θέμα της αξιοπιστίας τώρα. Εδώ τα έχω περισσότερο με τα κράτη-μέλη, τα οποία έχουν μια στάση κάπως υποκριτική. Ορισμένες από αυτές τις χώρες εποφελούνται από την αφησιμία που υπάρχει για το ποιος είναι καθαρός εισφορές και όχι. Ένας υπουργό λέει 20% πρέπει να πηγαίνει από την αναπτυξιακή βοήθεια στις κλιματικές αλλαγές. Όχι, δεν συμφωνούμε. Αυτό που πρέπει να επενδυθεί στην κλιματική αλλαγή πρέπει να έρθει από αλλού. Δεν πρέπει να χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της αναπτυξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς πάει. Χαθήκαν οι πόροι από την ανάπτυξη. Ας επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας λοιπόν στην αξιοπιστία του έργου μας και του λόγου μας. Σίγουρα υπάρχει η κρίση, υπάρχει η ανασφάλεια στον κόσμο. Άρα, ακόμα περισσότερο σημαντικό είναι να έχουμε στέρεα σημεία αναφοράς. Και αυτά υπάρχουν στη συνένεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανάπτυξη. Δεν σας εκπλήξει να επανέλθω σε αυτό το θέμα. Ελπίζω ότι η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα μπορέσει να συνυπογράψει το έγγραφο για την συνένεση όσον αφορά την ε, ανάπτυξη. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι τώρα μετά την κρίση να κάνουμε τα ίδια όπως και πριν της κρίσης. Δεν είναι σωστό αυτό, γιατί πρέπει να μείνουμε πιστοί στη δράση που προτείνει το έγγραφο αυτό. Και ετοιμάζω ένα ψήφισμα στο οποίο σας ζητάω να συνυπογράψετε αυτό το αγγραφό. Και τέλος, θα είμαι κάπως ομός, αυτοί που έχουν κάτι να προσφέρουν στην αξιοπιστία της ενωσιακής πολιτικής για την ανάπτυξη, να εμφανιστούν χώρες όπως η Νορβηγία ή και άλλες. Αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες που στις επόμενες διεθνείς διασκέψεις θα πούνε πολλά, και η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι πρέπει να υιοθετήσει μια ιδιαίτερα φιλόδοξη στάση. Επειδή έχει κύρος, έχει εμπειρία, έχει πραγματογνωμοσύνη. Οι άλλοι ας φροντίσουν και να πούνε ό,τι έχουν να πούνε, αλλά να τα κάνουν και πράξη. Και όποιος μπορεί να προσφέρει ε, στην ανάπτυξη ανά τον κόσμο, ας το κάνει, ας εμφανιστεί. Και εγώ έχω να ρωτήσω μερικά πράγματα τη λέει Διάστον. Πρώτον, μία διαπίστωση. Η συμμετοχή των κρατών μελών στην αναπτυξιακή βοήθεια ήταν 0,44% του ΕΠ το 2010, 0,42% το 2011 και 0,39% το 2012. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο κρίσης. Η ανθρωπιστική βοήθεια που είναι τόσο αναγκαία, δυστυχώς υποφέρει περισσότερο. Και εδώ υπενθυμίζω την περίπτωση της Συρίας. 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες που θα γίνουν 3 εκατομμύρια μέχρι τα τέλη της χρονιάς. 1 εκατομμύριο πρόσφυγες στην Ιορδανία. Επίσης Βόρειο Ιράκ, Λίβανος. Όλα τα μέσα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε ενώ τα χρήματα μειώνονται. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Άστον, εσείς τι δράσεις θα αναλάβετε για να πείσετε τους εταίρους μας, αυτούς για παράδειγμα που δεν αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες όπως η Γερμανία, να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και να φτάσουν στο 0,7% που έχουν υποσχεθεί. Δεύτερο σημείο. Η Επιτροπή μα ανησυχεί ιδιαίτερα για την τεχνική του συνδυασμού χρηματοδοτήσεων που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε την ανεπάρκεια δανείων. Το blending αυτό όμως οδηγεί σε χρέωση. Κάνετε ώστε η βοήθεια αυτή να μην καταλήξει σε υπερχρέωση την οποία να μην μπορούν να αντέξουν οι πιο φτωχές χώρες. Τρίτο, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο θέμα της συνοχής των πολιτικών μας, εξωτερικής, αναπτυξιακής, ασφάλειας. Βλέπουμε το πρόβλημα με διάφορα παραδείγματα. Μαλή, για παράδειγμα. Η κατάσταση οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στην υποανάπτυξη του Μαλή. Το Μαλή είναι μία από τις χώρες νοτίως του Σαχέλ αποσταθεροποιημένη. Η αναπτυξιακή βοήθεια λοιπόν έχει τεράστια σημασία για αυτή τη χώρα. Είναι όμως και θεμελιώδου σημασία για την ασφάλεια της Ευρώπης και τη περιοχή αυτή βέβαια. Υπάρχει και η Δυτική Σαχάρα στην περιοχή. Εσείς πώς θα βοηθήσετε. Η αναπτυξιακή βοήθεια θέλω να πω ότι είναι παράγοντας ασφάλειας. Το βλέπουμε και στο Αφγανιστάν. Εσείς θέλετε να κρατήσετε ε, στο επίπεδο των 200 εκατομμυρίων. Αυτό είναι καλό. Λοιπόν, ρωτάω, έχετε και εσείς τις ίδιες ανησυχίες με εμένα για τη διαφθορά στο Αφγανιστάν. Γίνεται κάποια έρευνα για την τράπεζα της Καμπούλ που έδειξε ότι 900 εκατομμύρια ευρώ, πέντε έτη αναπτυξιακής βοήθειας δηλαδή, τα καταχράστηκαν κάποια άτομα και ότι από αυτά τα 950 εκατομμύρια, 450 εκατομμύρια πήγαν στο Ντουμπάι, που είναι ε, φορολογικός παράδεισος. Και φάνηκε αυτό από την έρευνα που έκαναν οι ίδιοι Αφγανοί. Ε, με τα χρήματα που χρησιμοποιούν για να ενισχύσουν τους θεσμούς τους. Αυτή τη φορά δούλεψε το σύστημα γιατί οι δικαστικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τα χρήματα αυτά στο Ντουμπάι. Το Ντουμπάι όμως εξακολουθεί να είναι φορολογικός παράδεισος αδιάβατος. Αυτά είναι παραδείγματα που δείχνουν ότι η προβληματική των φορολογικών παραδείσων είναι άρρηκτα συνδυασμένη με την αναπτυξιακή βοήθεια και ότι αν δεν επιτεθούμε σε αυτό το φαινόμενο δεν θα προχωρήσουμε ούτε στο Μαλί ούτε στο Αφγανιστάν. Συνεπώς η ερώτησή μου είναι τι μέτρα σκοπεύετε να αναλάβετε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν καταφέρει να συμφωνήσει με μηχανισμούς τόσο βασικούς όπως είναι η ανταλλαγή πληροφοριών στο εσωτερικό της. Για να καταπολεμήσουμε τους φορολογικούς παραδείσους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στα πλαίσια του G20 ή του G8 που θα έπρεπε να αποτελεί στοιχείο της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Συνοχή σημαίνει να λύσουμε και τις διαμάχες που υπάρχουν και να δώσουμε και να μην δώσουμε προνόμια στη Μιαμάρ όσο παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και διώκει τη μουσουλμανική κοινότητα. Οπότε ρωτάω τι θα κάνετε για να σταματήσει η δίωξη αυτή της μουσουλμανικής μειονότητας στη Μιαμάρ. <clears throat> Έχετε το λόγο κυρία στον για να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Και μετά θα περάσουμε σε δεύτερο γύρο ερωτήσεων, έτσι. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Κύριε Μίτσελ, εσείς θέσατε τρεις ερωτήσεις, ε, νομίζω. Καταρχήν, η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το εμπάργκο όπλων. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι δεν ε, παρέχουμε όπλα ως ε, θεσμός. Το Συμβούλιο χθες το βράδυ κάθισε μέχρι πολύ αργά για να σκεφτεί πώς μπορεί να στηρίξει με τον καλύτερο τρόπο τους ανθρώπους της Συρίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφασίσει κανείς ποια μηνύματα θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο και το Συμβούλιο, όπως είδατε, αποφάσισε να παράσχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε απόφαση ε, που θα ληφθεί θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο. Αλλά η Ευρω... Ε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν συμμετέχουν. Έχετε δίκιο ότι η μείωση των επιπτώσεων των καταστροφών είναι πολύ σημαντικό θέμα και βέβαια έχουμε προγράμματα με τα οποία εξετάζουμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε τις χώρες ώστε να τις βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις καθώς και να προλάβουν κρίσεις. Αυτά τα κάνουμε με διάφορους τρόπους, αλλά να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Καταρχήν με τη συνεργασία με διάφορες χώρες, ε, ώστε να μπορούμε να δούμε πώς μπορούν να υπολογίσουν τις πιθανότητες ε, και τον αντίκτυπο μιας φυσικής καταστροφής. Ε, για παράδειγμα, σε μια... μπορεί να έχουμε κάποια περιοχή όπου να έχει συμβεί μια σειρά καταστροφών ε, είχαμε ένα τέτοιο πρόγραμμα στη Βυρμανία, τώρα συνομιλούμε με την Ινδονησία, έχουμε σε διάφορα μέρη του κόσμου. Το άλλο θέμα είναι να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να αναπτύξουμε μία ε, αίθουσα κινδύνου, να την πούμε έτσι, ώστε να μπορούν ε, να ανταποκρίνονται γρήγορα, ώστε να μπορούν να σώσουν όσο γίνεται περισσότερες ζωές σε περίπτωση καταστροφής. Από τη μία δηλαδή θέλουμε να μειώσουμε την πιθανότητα να συμβούν καταστροφές και από την άλλη θέλουμε να βοηθήσουμε στην ε, αντιμετώπιση των καταστροφών εφόσον συμβούν. Είχατε δίκιο όσον αφορά την ε, εξοικονόμηση χρημάτων, ε, είχατε επίσης δίκιο όσον αφορά τις ζωές που μπορούμε να σώσουμε. Τι γίνεται με τα κορίτσια. Ε, πριν πολλά χρόνια συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα για την για να βοηθήσουμε να αναγνωριστεί η αξία των ε, γυναικών και των κοριτσιών, η αξία ε, των γυναικών και των κοριτσιών στην κοινωνία. Και εμείς θέλουμε να ε, να δείξουμε την σημασία των κορισιών και των γυναικών στις κοινωνίες. Γι' αυτό επικεντρωνόμαστε στο ρόλο των γυναικών και στις ζωές των γυναικών και κοριτσιών. Ε, αυτό δεν αφορά μόνο την εκπαίδευση, έχει να κάνει ε, και με την αίσθηση του κόσμου ότι οι γυναίκες παίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινότητά τους, αλλά ότι επίσης είναι στοιχείο κλειδί και ίσο ε, μέρος της κοινωνίας. Θέλουμε λοιπόν, ε, και ε, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο ώστε να περάσουν οι ιδέες αυτές ε, στις κοινότητες. Αυτός είναι ο πυρήνας της αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού σε χώρες όπου δυστυχώς βλέπουμε ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια απαξιούνται. Κύριε Κορτέστε Λάστρα, με ρωτήσατε σχετικά νομίζω με την αναθεώρηση που κάνουμε. Ο στόχος είναι να δούμε τι λειτουργεί καλά και τι μπορεί να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα και να προσπαθήσουμε, όπως είπατε, να βρούμε τρόπους ε, να ενεργούμε καλύτερα μαζί, να συνεργαζόμαστε καλύτερα. Το θέμα λοιπόν είναι όχι μόνο μεταρρύθμιση ε, της ε, υπηρεσίας μας, αλλά και του τρόπου που εργαζόμαστε. Και ε, η συμβολή του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντική στο θέμα αυτό. Ο τρόπος εργασίας μας δεν είναι τέλειος, πρέπει να βρούμε τρόπο να τον βελτιώσουμε. Επίσης αναφερθήκατε στη συνέπεια των πολιτικών και την οριζόντια φύση των διάφορων πολιτικών. Σύμφωνο μαζί σας. Ένα από τα βασικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και είναι κάτι το οποίο ε, πιστεύω εδώ και πολύ καιρό, ε, αλλά βλέπω τρόπο να βελτιώσουμε ε, την κατάσταση είναι εξετάζοντας τον αντίκτυπο των πολιτικών, μα ε, μας μεταξύ τους. η συνέπεια, η συνοχή στην πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι δεν είναι αδύνατο να σκεφτούμε κάποια περίπτωση όπου μία πολιτική ουσιαστικά είναι καταστροφική για πολιτική σε έναν άλλον τομέα. Εάν δεν είμαστε προσεκτικοί λοιπόν και αν δεν δούμε τι άλλο κάνουμε, τότε μπορεί οι αναπτυξιακές πολιτικέ μας να είναι λιγότερο αποτελεσματικέ ε, από ό,τι θέλουμε. Ε, όταν λοιπόν σκεφτόμαστε η, εξωτε... η υπηρεσία εξωτερική δράση ε, πώς λειτουργεί, πώ μπορούμε να στηρίξουμε τις ε, τοπικές κοινότητες ε, και κοινωνίες προσπαθούμε ε, να εξετάζουμε το πλήρες φάσμα των πολιτικών, ε, την εκπαίδευση και την υποστήριξη παιδιών, προγράμματα που να βοηθούν τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις πολιτικές τους, υποστήριξη για ξεκίνημα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ειρήνη και ασφάλεια που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους, στήριξη για το, για το κράτος δικαίου, ανάπτυξη των διαφόρων θεσμών και καταπολέμηση τις διαφθορές. Όλες αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να συνδυάζονται σωστά μεταξύ τους ε, για να ε, είναι αποτελεσματικές και πιστεύω ότι στον τομέα αυτών μπορούμε να ε, βελτιώσουμε τον τρόπο εργασίας μας. Για παράδειγμα, ε, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος ε, μας μίλησε για τι γίνεται μετά το Ρίο, για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις διάφορες πολιτικές. Ε, επίσης, η επικοινωνία είναι ζωτική σημασία, είναι μία από τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το πώς μπορούμε να δείξουμε, να μεταφέρουμε το μήνυμα σχετικά με το τι κάνουμε. Στην ανθρωπιστική βοήθεια, ότι είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής του κόσμου, ότι είμαστε ο σημαντικότερος υποστηρικτής ε, των ε, Ηνωμένων Εθνών και τα Ηνωμένα Εθνή το λένε αυτό συχνά. Ε, πρέπει να δείξουμε, να διαφημίσουμε τι κάνουμε, διότι θυμηθείτε ότι πολλοί από την υποστήριξη μας είναι χρήματα που πηγαίνουν στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να κάνουν τη δουλειά που θέλουμε και έτσι παίρνουν όλη τη δόξα κατανοητό αυτό, αλλά πρέπει και εμείς να δείξουμε τι κάνουμε. Ε, κάποια κράτη-μέλη έχουν επιλέξει εντός του πλαισίου ε, να ε, ε, αποδώσουν το 20% των πόνων τους στην αλλαγή του κλίματος. Για το θέμα αυτό θα πω ότι η τελευταία φορά που μέτρησα περίπου 101 χώρες στον κόσμο μπορεί να επηρεαστούν δραματικά από την αλλαγή του κλίματος πολύ περισσότερο από ό,τι θα πληγούν, για παράδειγμα, χώρες ε, της ευρωπαϊκή Ένωσης. Μπορεί να δούμε ξηρασία, ε, πείνα, ε, πλημμύρες, αλλαγές που δεν μπορεί να υποστηρίξει η υποδομή της χώρας. Είδαμε τρομερές πλημμύρες τα τελευταία δύο-τρία χρόνια σε περιοχές λοιπόν, λοιπόν όπου είναι πιθανό να ξανασυμβούν τέτοιες πλημμύρες, αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις για τις κοινότητες αυτές. Το ίδιο ισχύει για τις περιόδους ξηρασίας. Εάν βρίσκεται κανείς σε μια κοινωνία όπου ο κόσμος ε, καλλιεργεί τα δικά του τρόφιμα, είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει εάν δεν βρει τρόπο να παρέχει νερό το οποίο είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης ε, της αλλαγής του κλίματος. Ε, είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζει κανείς τι θα γίνει με τις κοινότητες αυτές. Πολλές ε, τέτοιες κοινότητες εξαφανίζονται διότι ο κόσμος αναγκάζεται να μετακομίσει, διότι δεν μπορεί πια να ζει εκεί που θέλει να ζει. Αυτό επηρεάζει τις οικογένειες, επηρεάζει τα παιδιά και επηρεάζει την οικονομική βιωσιμότητα πληθυσμιακών ομάδων. Όταν λοιπόν σκέφτομαι την ε, ανάπτυξη και την αλλαγή του κλίματο, θεωρώ ότι τα δύο αυτά συνδέονται πάρα πολύ στενά μεταξύ του. Εάν δεν έχουμε συνείδηση ότι σε κάποιε χώρε ε, οι επιπτώσει τη ε, αλλαγή του κλίματο θα έχει δραματικέ επιπτώσει στι ζωέ των ανθρώπων, θα πρέπει να σκεφτούμε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για να στηρίξουμε την βιωσιμότητα των κοινοτήτων αυτών σε όλε τι περιπτώσει. Αν δεν το κάνουμε λοιπόν αυτό, είναι κάτι το οποίο θα μετανιώσουμε, διότι έχει να κάνει με την ε, όλη συνέπεια και συνοχή. Θα πρέπει να δούμε τις επιπτώσεις στους διάφορους τομείς πολιτικής. Ε, Όσον αφορά την ε, συνένεση για την ανάπτυξη, ε, ο λόγος που δεν τον έχω ε, υπογράψει είναι ότι καλύπτομαι, διότι είμαι πρόεδρος του Συμβουλίου. Δεν είναι επειδή δεν έχω επιθυμία, επειδή δεν θέλω να υπογράψω, αλλά δεν χρειάζεται. Αλλά εάν αυτό σας οικονοποιεί, για μένα δεν είναι θέμα, εάν είναι να σας ικονοποιήσω να υπογράψω. Αλλά ε, σας παρακαλώ μην ερμηνεύσετε τη μη υπογραφή ως ε, έλλειψη βούλησης. Απλά κάθε φορά που το έλεγξα και το, το ξανάλεξα και σήμερα, ε, οι νομικοί μου λένε ότι καλύπτεστε κατά 100% από το έγγραφο αυτό. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε λοιπόν. Παρακαλώ μην θεωρήσετε ότι ότι είναι έλλειψη βούλησης. Και κυρία Ζολή, έχετε δίκιο. Ε, τα νούμερα δείχνουν ε, το, ε, ότι μειώνεται το ποσοστό ε, των ε, πόρων που δίνουμε και οι δύσκολες καταστάσεις μας αναγκάζουν να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία και εντός και εκτός της χώρας στους ε, Σύριους εντός και εκτός της χώρας. Ε, επισκέφτηκα ε, τα στρατόπεδα προσφύγων στη Γιορδανία. Είμαστε σε συνεχή επαφή μέσω των αντιπροσωπιών μας. Είναι τρομερή κατάσταση. 100 εκατομμύρια ευρώ έχουμε δώσει μέχρι τώρα αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν ε, τελειώσει αυτή η τρομερή τραγωδία θα πρέπει να ανοικοδομηθεί μια χώρα, θα, θα, θα πρέπει να επιστρέψει ο κόσμος να βρει σχολεία, δρόμους, ε, κατοικίες. Ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε ένα έθνος το οποίο ε, θα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και πολλοί κόσμος θα έχει τραυματιστεί από τις εμπειρίες αυτές. Όλα αυτά θα απαιτήσουν πολλά χρήματα, διότι ε, τα χρήματα θα είναι στοιχείο κλειδί σε όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση και το κάνουμε αυτό ε, σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να πούμε ότι η δεσμεύσει σας εδώ είναι επένδυση, δεν χαρίζουμε χρήματα, πρόκειται για επένδυση για το μέλλον των δικών σας ανθρώπων και των δικών σας κοινοτήτων, διότι τον έχουμε οι ισχυρές αναπτυσσόμενες ε, χώρες ε, είναι χώρες που, ε, με τις οποίες κάποια μέρα θα έχουμε εμπορικέ σχέσεις, θα τις επισκεφτούμε, θα είμαστε τουρίστες εκεί, ενώ οι χώρες που καταραίουν θα συναντήσουν δυσκολίες με τις οποίες θα πρέπει να ασχοληθούμε. Πρόκειται λοιπόν για επένδυση στο μέλλον των δικών μας ανθρώπων αλλά και των ε, χωρών αυτών. Ε, αυτό είναι το ε, μήνυμα που θέλω να στείλω. Όσον αφορά το συνδυασμό επιχορηγήσεων και δανείων, αυτό είναι σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είχα αρκετές εμπειρίες στο θέμα αυτό. Πρέπει να προσέξετε να το κάνετε αυτό με τρόπο τέτοιο που να μην δημιουργεί υπερβολικό χρέο για χώρε που δεν μπορούν να το ε, αποπληρώσουν. Μπορεί να χρησιμοποιήσει κανεί όμω με δημιουργικό τρόπο τα χρήματα, του πόρου. Ε, και τα τελευταία δύο χρόνια ιδιαίτερα θεωρώ ότι πρέπει να ε, φερθούμε πιο έξυπνα. η δουλειά λοιπόν που έχουμε κάνει στην Τινησία, τη Ιορδανία, στην Αίγυπτο και που θα κάνουμε στη Βυρμανία, Μιανμάρ, είναι να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε διάφορου πόρου ώστε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Όχι να δημιουργήσουμε χρέη, αλλά να παράσουμε ε, με υποστήριξη με δάνεια με ευνοϊκούς όρους, ε, με χορηγίες ε, δεν θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια κατάσταση επιβλαβή για τις χώρες αυτές. Ε, θέλουμε απλά να πετύχουμε πιο αποτελεσματική χρήση ε, των πόρων. Και κυρία Ζολή, έχετε δίκιο όσον αφορά ε, την συνοχή. Το Μαλί είναι πολύ καλό παράδειγμα. Η στρατηγική μας για τη ζώνη Σαχέλ στόχο έχει να εξετάσει όλες τις ανάγκες της περιοχής. Ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα, νερά, εκπαίδευση, υποστήριξη για υπηρεσίες υγείας. Είναι ε, πολύ δύσκολο το θέμα της ειρήνης και ασφάλειας σε μια χώρα με ε, μη σταθερά σύνορα. Ε, η στρατηγική μας λοιπόν για τη ζώνη Σαχέλ μας ανάκασε να το σκεφτούμε ε, αυτό. Και όσον αφορά το χρήμα και πού θα πάει, το να παρακολουθεί κανεί τη ροή των χρημάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα από τα θέματα ε, με τα οποία ασχοληθήκαμε στην ε, Σομαλία είναι να δούμε πού πάνε τα χρήματα, τα έσοδα από την πειρατεία, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτού που λαμβάνουν τελικά τα χρήματα αυτά. Το ίδιο ισχύει για τη διαφθορά. Και ξέρω ότι υπάρχουν πολλέ πρωτοβουλίε. Η Κομισιόν έχει ασχοληθεί με διάφορε πτυχέ. Το G8 σίγουρα θα, το G8 σίγουρα θα το συζητήσει αυτό. θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Ε, ε, πάντως, ε, ένα από τα θέματα για τη Βυρμανία ένας από τους τομείς με τους οποίους θα ασχοληθούμε είναι η εκπαίδευση της αστυνομίας, διότι ένα από τα προβλήματα είναι η ανικανότητα των τοπικών δυνάμεων να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις και να διαφυλάσσουν την ηρεμία. Ε, πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τις χώρες ε, να αντιμετωπίζουν ε, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε τώρα ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων για την κυρία Άστον, ο κύριος Κασμαρέκ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Άστον, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω γιατί αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Σήμερα έχω την αίσθηση ε, ότι ε, είμαι μέλος του γραφείου σας ε, και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω φόρτου εργασίας να αποδεχτείτε προσκλήσεις. Έχετε και την Ολομέλεια της Euronest, όπου νομίζω ότι είχατε επίσης προσκληθεί. Ε, γι' αυτό λοιπόν ειλικρινά σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την ε, πρόσκλησή μας. Ξέρω ότι αυτές οι επιλογές είναι πολύ δύσκολες. Δεύτερον, να σας ευχαριστήσω για όσα είπατε και για όσα πράτετε. Όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια, είμαστε πολύ περήφανοι. Σήμερα είδαμε τον κατάλογο των δωρητών και ε, με περηφάνεια βλέπουμε ότι είμαστε επικεφαλής. Όμως από την ε, άλλη πλευρά μονάχα τέσσερις χώρες μέλη, η Σουηδία, η Δανία, το Λουξεμβούργο ε, και η Μεγάλη Βρετανία έχουν καλύψει πλήρως τις υποσχέσεις δεσμεύσεις τους. Στην, στον, του καταλόγου είναι οι χώρες οι οποίες δίνουν το 0,08% ε, του ΑΕΠ σε αναπτυξιακή βοήθεια, δηλαδή 8 φορές λιγότερο από ό,τι θα έπρεπε. Πρέπει να μας στηρίξετε εδώ στην Επιτροπή μας, γιατί συχνά ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά και εκ των προτέρων σας ευχαριστώ ε, για την πίεση που σίγουρα θα ασκήσετε στους υπουργούς εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνετε αυτό. Ερώτηση τώρα. Για να αξιολογήσουμε την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει οπωσδήποτε να αναλυφθούν περαιτέρω δράσεις ε, αλλά αναλογιζόμενοι όλο αυτό το πλαίσιο, το πιο δύσκολο ε, στην ανάλυση είναι να αναλύσουμε τον στόχο 8, δηλαδή την ατζέντα μετά το 2015. Υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν οράματα, έτσι ώστε ε, αυτές οι σφαιρικές συνολικές ε, εταιρικέ σχέσεις να επιτευχθούν, γιατί κατά την άποψή μου αυτός θα είναι ο πιο δύσκολος στόχος στην επιτευχή στην επίτευξή του. Αλλά πρόκειται και το μέλλον μας, άρα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, να ενεργήσουμε γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε της χιλιτίας σας είναι ιδιαίτερος προσφυλής και όπως ξέρετε λαμβάνει η χώρα μια πολύ σημαντική συζήτηση σχετικά με τους επόμενους στόχους της χιλιετίας. Αυτή η ιστορία ε, του, της χιλιετίας ήταν ε, μια επιτυχημένη ιστορία, ένα success story. Και ο στόχος ε, της καταπολέμησης της ένδυας δεν ολοκληρώθηκε το 2015 αλλά το 8. Ξεκινάει τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα πιο φιλόδοξο στόχο που θα μπορούσε να είναι ε, η κατάργηση της απόλυτης φτώχειας στα επόμενα 15 χρόνια. Μια συζήτηση η οποία βεβαίως ε, εμπλέκει πολλούς εμπειρογνώμονες και τα μεγαλύτερα ιδρύματα, θεσμικά, θεσμικές υπηρεσίες κτλ. Ποια είναι η άποψή σας, τι θα μπορούσε να δώσει, ε, τι θα μπορούσε, πώς θα μπορούσε να συμβάλλει σε αυτόν τον ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Νιούτον Ντάν. Και εγώ μια ε, σύντομη ερώτηση. Η κυρία Ζολία ανέφερε στην ερώτησή της το Ντουμπάι. Ε, εγώ ασχολούμαι με την Επιτροπή για το Οργανωμένο Έγκλημα ε, και στο Ντουμπάι συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Η, Ευρώπη πλημμυρίζει από παραχαραγμένα προϊόντα, προϊόντα απομίμησης, αλλά η, το, το Ντουμπάι οποτεδήποτε οποτεδήποτε ε, ε, πιάνουν ας πούμε τέτοια προϊόντα ε, αντί να τα κατασχέσουν όπως γίνεται συνήθως τα στέλνουν πίσω και να τα καταστρέψουν, τα στέλνουν πίσω στο κατασκευαστή έτσι ώστε να ψάξει να βρει μια άλλη οδό για να προωθήσει τα προϊόντα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το ε, δούμε, με ποιο τρόπο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Την, ε, σε ένα χρόνο επίσης, όπως ξέρετε, αλλάζει το κοινοβούλιο, ε, έχουμε εκλογές ε, και βεβαίως ε, ίσως να μην ξανάρθετε μέχρι τότε και ίσως όταν θα ξανάρθετε να μην είναι οι ίδιοι βουλευτές, αλλά βεβαίως αυτό δεν είναι κανονική ερώτηση. Η κυρία Τόγια παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και από τη δική μου πλευρά. Νομίζω ότι ίσως ε, να έρθετε ακόμα πιο πολύ και πιο σύντομα να σας έχουμε κοντά μας λόγω ακριβώς των εκλογών. Εν πάση περιπτώσει, ε, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επαφές με σας και με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης της οποίας, είστε, της υγείστε, έτσι ώστε να μιλάει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε εξωτερικό επίπεδο με μία φωνή. Είναι δύσκολη η δουλειά σα, αλλά σα στηρίζουμε παρόλα αυτά. Δύο ερωτήσει, μία πιο απλή, μία λίγο πιο δύσκολη, αλλά κατά την άποψή μου σημαντική. Πρώτη ερώτηση. Στην συζήτηση για του στόχου ε, μετά το 2015 διαφαίνεται όλο και περισσότερο, αναδύεται όλο και περισσότερο και στην Επιτροπή μας εδώ ε, η ανάγκη να υπάρξουν οι σωστοί στόχοι αλλά και η κατάλληλη μεθοδολογία έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως επιτυγχάνονται αλλά με μεγάλο ξόδεμα δυνάμεων, πόρων κτλ. Επίσης, ποιος είναι, ποια είναι η διάρκεια των στόχων ε, αυτών τα κριτήρια αξιολόγησης οπωσδήποτε συνδέονται με τη σταθερότητα, με την, ε, με την ε, διάρκεια στο χρόνο κτλ. Επομένως, η, η ικανότητα να ενστερνίζει κανείς τα αποτελέσματα, η ικανότητα ε, να εμπεδοθούν τα αποτελέσματα και βεβαίως η επίτευξη των στόχων αλλά και η ταυτοποίηση των ιδίων και αυτό πάντα έγινε ε, μέσα από την ε, ε, μέσα και από συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών που είναι αυτό το δυνατό, ισχυρό, υγιές τμήμα της κοινωνίας που πάντα είχαμε στο πλευρό μας. Επίσης το θέμα της διαφθοράς είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά παντού. Πώς λοιπόν μπορούμε πέρα από τα σλόγγαν και πέρα από τα, ε, από τα ε, πολιτικά έτσι, μηνύματα και τις επικεφαλίδες, πώς μπορούμε ε, να σταθεροποιήσουμε τη σχέση με την κοινωνία των πολιτών. Δεύτερη ερώτηση, πιο περίπλοκη, ποιο, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, ποιο είναι το πρόγραμμα από τη δική σας πλευρά έτσι ώστε ε, να συμβάλλεται εις ε, την ανάπτυξη ε, του διεθνούς δικαίου. Βεβαίως με συνεργασία, με με τις δωρεές, με τις δεσμεύσεις ε, και ε, βεβαίως ε, εδώ θα ήθελα να στιγματίσετε και τη δικιά μου χώρα εάν δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της γιατί όπως είπε και η πρόεδρος Ζολή από το 0,44 φτάσαμε στο 0,41 και τώρα στο 0,39 για το 2012. Μιλάμε για το διεθνές δίκαιο. Ποιος το προωθεί το διεθνές δίκαιο. Αλλά στην ουσία και στην Οτάβα ας πούμε η κοινωνία των πολιτών κινήθηκε στη Γενέβη το ίδιο όταν αρχίσουμε ε, να ε, μιλάμε, ε, όταν ας πούμε στη Γενέβη ξεκίνησε η συζήτηση ε, για την, ε, για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού, ήδη είχε ήδη ξεκινήσει η συζήτηση στην κοινωνία των πολιτών. Όταν μιλάμε τώρα για το land grabbing, όταν μιλάμε επίσης για κανόνες διεθνείς που είναι μονομερείς, γιατί δεν είναι οι σοβαροί αυτοί οι κανόνες και οι και βεβαίως ε, το θέμα της γης ε, εμπλέκεται και με άλλα ζητήματα. Είναι με το θέμα της διατροφής, των τροφίμων και επομένως πρέπει να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις. Κατά την άποψή μου ε, γίνονται κάποια βήματα στα πλαίσια της Ένωσης της Αφρικής, αλλά θα πρέπει ε, ή το Ηνωμένα Έθνη ή κάπου αλλού ε, να ξεκινήσει, να ενστερνιστούν οι διάφορες, οι διάφορες ε, θέσεις αυτές, να τις ασθενιστούν ε, οι υπηρεσίες. Πώς μπορείτε να κάνετε εσείς να πάρετε μέρος ε, σε, αυτές, σε αυτούς τους αγώνες για να προωθήσετε το Διεθνές Δίκαιο. Ευχαριστώ πολύ. Ακόμα ένας ομιλητής ζητάει το λόγο. Θα είναι η τελευταία ερώτηση και μετά θα ζητήσουμε την Λέδη Άστον να απαντήσει και να ολοκληρώσει. Κύριε Γκέρενς, έχετε το λόγο για την τελευταία ερώτηση. η ύπατος εκπρόσωπος δεν θα εκπλαγεί αν δει ότι επιμένω στην διεκδικησή ε, μου, δηλαδή που θέλω να σας δω να υπογράφετε το κείμενο για την ανάπτυξη. Και έχω και άλλα τρία επιχειρήματα. Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία. Δεύτερο επιχείρημα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το υπέγραψε το κείμενο γιατί πιστεύουμε ότι όλοι οι θεσμοί πρέπει να αναγνωρίσουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο για την αναπτυξιακή συνεργασία. Τρίτον, δεν ξέρω αν αυτό θα σας ε, πείσει, αλλά το Λιράνος είπε ότι αν εννοείται, χωρίς να το πούμε, καλύτερα να το πούμε. Και εγώ θα έλεγα, αν ισχύει χωρίς να το υπογράψετε, ε, ακόμα καλύτερα θα είναι αν το υπογράψετε. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι αν μπορούμε να βρούμε μια ημερομηνία και μια τελετή για την υπογραφή, θα έρθουμε πολύ άριθμοι μαζί σας για να σας χειροκροτήσουμε με επιμονή. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Άστον, έχετε το λόγο για να απαντήσετε και να ολοκληρώσουμε έτσι το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα εξηγήσω, με τον, θα εξηγήσω τον κύριο Κάσμαρεκ και να σας πω ότι περιμένουμε την έκθεσή σας. Έχετε δίκιο Υπάρχουν πολλές συναντήσεις και συνέχεια πρέπει να κάνω μια επιλογή, αλλά χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Συνεχίζουμε να πιέζουμε τις χώρες προκειμένου να φέρουν σε πέρα στις υποχρώσεις τους. Και είναι δύσκολο. Ένα από τα θέματα είναι πώς μπορείς να εξηγήσει στον κόσμο, στο κοινό σου, ότι αξίζει τον κόπο να πάνε αυτά τα χρήματα στην ανάπτυξη. Σε ορισμένε χώρε αυτό δεν γίνεται καλά και υπάρχει πρόβλημα. Άρα πρέπει να βρούμε και τον τρόπο να τους βοηθήσουμε να περάσουν αυτό το μήνυμα ότι πρόκειται για μια επένδυση η οποία θα μας αποφέρει, θα αποφέρει στις χώρες εκείνες οι οποίες ε, δίνουν τα χρήματα αυτά στην ανάπτυξη γιατί ε, είναι μια επένδυση. Επιπλέον υπάρχει και το ηθικό επιχείρημα ότι βοηθάμε τον κόσμο να μην πεθαίνει. Όμως χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά για να περάσει το μήνυμα αυτό ότι πρόκειται για μια επένδυση. Εμείς λέμε ότι είναι κάτι που όλοι συμμεριζόμαστε. Πρόκειται για μια αξία. Τώρα, ένα από τα πράγματα που συζητήσαμε σήμερα είναι να μπορέσουμε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο να συμφωνήσει για το προς τα που πάμε κράτος δικαίου, δημοκρατική διακυβέρνηση και λοιπόν όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αυτό που βγήκε πάντως ξεκάθαρα από τη ζήτηση με τα κράτη-μέλη και από τη συζήτηση που είχαμε με τα Ηνωμένα Έθνη είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερη συνδυτοποίηση για το ότι πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί κατά της διαφθοράς, ερικοδόμηση θεσμών. Έτσι φτιάχνετε μια κοινωνία όταν έχει τις υποδομές που χρειάζεται και τότε μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Ε, κύριε Λάκη, δεν ήμουν σίγουρη ότι ήσασταν εδώ. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω. Αυτό που λέτε για την απάλληψη της ένδυας, ε, σίγουρα είναι σημαντικό. Στο πάνελ υψηλού επίπεδου συζητιέται για μετά το 2015 πώς θα συνεχίσουμε με το στόχο αυτό απάλληψη της ε, πλήρους φτώχειας. Βέβαια, η ε, επικεφαλής εκεί θα ήταν ε, περισσότερο σε θέση να σας απαντήσει παρά εγώ. Πάντως κάνει πολύ καλή δουλειά. Τώρα το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Πέρα από το να βγάλουμε τον κόσμο από την απόλυτη ένδια, πρέπει να δούμε και πώς θα βοηθήσουμε τον κόσμο αυτό να παραμείνει εκτός της απόλυτης άδεια. Και πέρα από τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε συνέχεια και τους κινδύνους που ελοχεύουν, υπάρχουν χώρες όπου ξέρουμε ότι έχουν πάρα πολλούς πόρους, πολύ πλούτο, αλλά δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν γιατί είναι σε πόλεμη κατάσταση. Είναι και αυτό ένα λόγο για τον οποίο δυσκολεύεται ο κόσμο να βγει από την ένδια. Έχουμε πολλά παραδείγματα όμως που έχουν αποδώσει και που δείχνουν ότι τελικά και με λίγους πόρους μπορείς να κάνεις φοβερά πράγματα για να βοηθήσεις τον κόσμο να βγει από τη φτώχεια. Και ο κόσμος ε, δράτη ό,τι του προσφέρεις για να αποφεληθεί και να βγει από τη φτώχεια. Για παράδειγμα, τι κάνουν οι γυναίκες, οι κοινότητες γυναικών, πώς φτιάχνουν επιχειρήσεις, πώς ε, βοηθούν τους υπόλοιπους. Είναι μεγάλη φιλοδοξία. Πρέπει να το κάνουμε. Είναι γελίο το 2013 να καθόμαστε και να παρατηρούμε διαφημίσεις από καταπληκτικές μη κυβερνητικές οργανώσεις που βοηθούν τον κόσμο που ζει όλη τη φτώχεια. Είναι τροπή να καθόμαστε στον καναπέ και να τα κοιτάμε. Και σας θέλω να σας ευχαριστήσω και την Ιντοντάν για αυτό που είπατε για το Ντουμπάι και για τις εκλογές. Ε, εντάξει, καλή τύχη στο κάτω-κάτω σε όλους. Αυτό έχω να σας ευγηθώ τώρα του χρόνου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πλησιάζουμε στις εκλογές. Θα είναι η στιγμή που θα έχει η Ευρώπη για να προβληματιστεί σε μερικές χώρες περισσότερο από αλλού, τέλος πάντων, δεν μπούμε σε λεπτομέρειες. Κυρία Τόγια, η κοινωνία των πολιτών είναι επικεφαλή στην κοινωνία. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι, όπως το περιγράφεται, εισπράττουν τα προβλήματα του κόσμου και μας ζητούν να τα δουλέψουμε και να υπογράψουμε διεθνείς συμφωνίες για να τα λύσουμε. Η κοινωνία των πολιτών ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή του μετόπου για τις τρομερές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στις κοινωνίες. Υπάρχουν χώρες που είναι σε μεταβατική κατάσταση. Εγώ θέλω να φροντίσω η κοινωνία των πολιτών να βρίσκεται στην καρδιά. Δηλαδή, να μην, δεν φτάνει να πηγαίνουν σε εκλογές οι χώρες και να έχουν εκλογές πρέπει η κοινωνία των πολιτών να μπορεί να συμμετέχει και μετά. Και όπου και πηγαίνω, στην Τινησία για παράδειγμα, όταν ε, μπαίνω σε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το λέω στον κόσμο που έχω συναντήσει, στη Λιβύη, στη Νιγηρία και έχω ακούσει τις ανησυχίες τους και την αποφασιστικότητά τους μέχρι τις κοινωνίες των πολιτών που ενισχύονται παντού στην Αφρική, στη Βερμανία, στο Αφγανιστάν. Υπάρχουν πραγματικές προσπάθειες που βοηθούν τον κόσμο να προδεύσει. Πρέπει να τους βοηθούμε και εκείνες μας βοηθούν πιέζοντάς μας για να πετύχουμε τους στόχους. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας. Και κύριε Γκέρελς, πώς μπορώ να αρνηθώ μια τόσο όμορφη πρόσκληση σαν και αυτή που μου κάνατε. Οπότε ναι, φυσικά, φυσικά. Αν αυτό θα σας κάνει ευτυχή βεβαίω. να οργανώσουμε μια τέτοια τελετή. Θα έχουμε και σαμπάνια. Να, σαμπάνια. Ωραία. Εντάξει, τέλο πάντων, οτιδήποτε. Για σας, με όλη μου την καρδιά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ωραία, με αυτά τα πολύ καλά νέα, ευχαριστούμε πολύ την Ήπατο εκπρόσωπο για την παρουσία της εδώ και για τις απαντήσεις που μας έδωσε. Σας ευχόμαστε πολύ κουράγιο για όλα αυτά τα καθήκοντα που έχετε να φέρετε σε πέρας. Βασιζόμαστε σε εσά προκειμένου να υποχρεώσετε τα κράτη-μέλη να φέρουν σε πέρα και αυτά τις υποχρεώσεις τους και να διασφαλίσουν μεγαλύτερη συνοχή στην εξωτερική μας πολιτική. Σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you. I'm leaving for Kabul oh. tomorrow morning. Oh, yes.